Καλημέρα, ξεκινήσουμε. Έχουμε ε, καλή απαρτία, έχουμε και κάποιους κοιόδης για το πρώτο σημείο. Για το πρώτο θέμα μας, καλωσορίζω θερμά τους παρισταμένους την πρώτη μέρα του διημέρου της συνεδριάσεως. Υιοθετείτε καταρχάς το σχέδιο μέσης διάταξης. Uh, uh, uh, Καλωσορίζω και το ακροατήριό μας που παρακολουθεί τη συνεδρίαση στο διαδίκτυο μέσω web streaming, όπως όλες οι συνεδριάσεις μάλωστε. Έχουμε και νέο έγγραφο της Επιτροπής που εκδίδεται πριν από τη συνεδρίαση, που πρέπει να το έχετε και στα γραφεία μοιράζεται των μελών για να τα δει στους επισκέπτες. Όποιος θέλει αντίγραφο, μπορεί να στείλει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που μας ακούει και σας στέλνουμε ηλεκτρονικά πριν από τη συνεδρίασή μας, σας στέλνουμε αυτό το έντυπο, τον ημερωτικό της Επιτροπής μας. Έχουμε κάποια πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων της 6ης Φεβρουαρίου και εκείνες θα θεωρηθούν, τα πρακτικά θα θεωρηθούν συγκεκριμένα εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις που θα υποβληθούν στη γραμματεία με το τέλος τη συνεδριάσεως της σημερινής. Πάμε στο πρώτο από τα βασικά θέματα της ημερήσιας διάταξης. Είναι αρκετά περίπλοκη η ημερήσια διάταξη, καλύπτει ευρύ φάσμα θεμάτων όλη την κλίμακα των εργασιών μας καλύπτει. Από την ενιαία αγορά αγαθών μέχρι άλλες τεχνικές προτάσεις. Ευρύτα το φάσμα. Ο Επίτροπος Σέμετα θα έρθει στις 11.30 στην Επιτροπή μας να μας μιλήσει για τα μελλοντικά σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τον τομέα τον φορολογικό και τον τελωνιακό και μετά έχουμε και μια σημαντική μελέτη για τον τελωνιακό κώδικα και θα μας μιλήσει ο κύριος Σέματα γι' αυτό. Αναθέσαμε σχετικά μια, συνταχθεί μια έκθεση. Θα με ενημερώσει και αυτό το θέμα, οπότε είναι καλό να παρίσταστε για να ακούσετε να μας πει. Πάμε στο πρώτο σημείο που είναι η έκθεση δική μου για την Επιτροπή μας όσον αφορά την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αναδιάθρωση της οδηγίας για τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη. Έγινε ανταλλαγή απόψεων όταν μας έκανε την παρουσίαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αξιολόγηση των συνεπειών της πρότασής της, συναντήθηκαν κοιότητες ηγητές και πήγαμε και σε αποστολή. Είδαμε αρκετά σκάφη στο Ντίσελντορφ. Συναντήσαμε διάφορου χρήστε των σκαφών αυτών και εκπρόσωπου βιομηχανία και θεώρησα ότι έχω αρκετέ πληροφορίε για να συντάξω μια έκθεση, η οποία σα παρουσιάζεται τώρα. Δεν θα αναφερθώ στις λεπτομέρειες όλες της εκθέσεως, διότι έχουν παρουσιαστεί προηγουμένως, αλλά θα ήθελα να σας κάνω με σύντομη παρουσίαση και να ακούσω σχόλια σκιωδών εισηγητών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. ορίζω την ομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρίσταται και θα συμμετάσχει στη συζήτηση. Ήταν μαζί μας στο ταξίδι που κάναμε στον σε αυτή η ομάδα της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής. Τα βασικά θέματα όσον αφορά την πρόταση ποια είναι. Δύο είναι αυτά. Πρώτα απ' όλα έπρεπε να επικαιροποιηθεί στις λεπτομέρειες η πρόταση. Είναι θεμητό να πούμε ότι η παρούσα πρόταση ε, λειτουργήσε όσο θα θέλαμε να λειτουργήσει μια οδηγία την αγορά για να δημιουργήσει μια νέα αγορά. Αλλά επειδή είναι αφήγηση σκαφών είναι παγκοσμίου μορφής ε, εγχείρημα ε, και είναι πολύ σημαντικός τομέας, ε, βέβαια είναι αυτό ο τομέα σχετικά μικρότερο όσον αφορά την αυτοκινητοβιομηχανία, σχέση με την αυτοκινητοβιομηχανία όσον αφορά τον όγκο παραγωμένων προϊόντων. Αλλά έπρεπε να εξετάσουμε και να σκεφτούμε τι κάνουμε όσον αφορά τον τομέα αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο, κάτι μα παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι έχοντα δει το φάσμα των σκαφών που προσφέρονται και συναντώντα διάφορου ναυπηγού που εξάγουν πολλά σκάφη σε όλο τον κόσμο και τα στέλνουν σε όλο τον κόσμο, είδαμε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ευθυγράμμιση με τους παγκόσμιους κανόνες. Όσον αφορά τις εκπομπές καυσαερίων, παραγωγή θορύβου και άλλες πτυχές που καλύπτει εν λόγω πρόταση. Όσον αφορά τις εκπομπές των εξατμίσεων, ε, νομίζω ότι η θέση μου είναι η εξής. Υποστηρίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ευθυγραμμιστούμε με τα παγκόσμια πρότυπα και αυτό προτείνω, με άλλα λόγια, να το αποδεχτούμε από την άλλη, νομίζω ότι είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι χρειάζεται ακόμα να γίνει η δουλειά, ούτω ώστε να ετοιμάσουμε τη νέα γενιά των ε, κινητήρων για τα πλοία, κυρίως για τα μικρά σκάφη και κυρίως τις εξολέμβιες μηχανές. Και από συζητήσεις με τους κατασκευαστές κινητήρων είδαμε ότι έχει ξεκινήσει αυτή η δουλειά, δηλαδή καταλαβαίνουν τις απαιτήσει που υπάρχουν να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι ήταν σημαντικό αυτή η πρόταση να αντικατοπτρίζει το ότι θα υπάρξει και άλλη φάση που θα ακολουθήσει. Δηλαδή θα είναι ένα κομμάτι μιας μεταβατική περίοδου. Και αυτό επίσης το έκανε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα μοτοποδήλατα που θα συζητήσουμε σε λίγο αργότερα. Αυτή είναι η πρότασή μου. Συνεπώς και θα ήθελα να ρίξουμε και μια ματιά σε κάποιες άλλες πτυχές οδηγίας, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι στο μέλλον ε, θα μπορεί να αποκριθεί στις καταστάσεις που μορφωθούν. Θα προβλέπει τις ενδεχόμενες αλλαγές. Ας πούμε αν έχουμε ε, υβριδικούς κινητήρες σε κάποια σκάφη και τα βιοκαύσιμα από όλο και περισσότερο θα χρησιμοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο. Και τη δυνατότητα επίσης να λάβουμε υπόψη τα βιοκαύσιμα. Όσον αφορά την παραγωγή θορύβου, θεώρησα ότι το θέμα του θορύβου καλύπτεται επαρκώς σχετικά με το τι μπορεί να επιτευχθεί μέσω νομοθεσίας. Το σκάφος ε, παράγει θόρυβο και από πλευράς κινητήρως και από πλευράς ε, ε, του μετακινήσεως του κήτους με ταχύτητα στη θάλασσα. Το, η πιο νέα εξέλιξη που έλαβε χώρα μετά τις πρώτες συζητήσεις με τους Κιώδης είναι το εξής. Έριξα εγώ μια ιδέα. Να εξετάσουμε τον ορισμό των κατηγοριών σχεδιασμού σκαφών. Αν δείτε τις κατηγορίες σχεδιασμού σκαφών στην πρόταση, καθορίζονται με βάση χρήση σκαφών που μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε ανοιχτή θάλασσα, παράκτια ή σε εσωτερική ναυσιπλοεία. Είμαι εγώ μηχανικός και από πλευράς μηχανικού πρέπει να πω ότι τα θέματα που καλύπτονται σχετίζουν και τις κλιματολογικές συνθήκες, το ύψος των κυμάτων και το γενικότερα το κλίμα. Ε, δηλαδή τους παράγοντες που πρέπει να λάβει υπόψη ο ναυπηγός για να αναφυγήσει ένα πλοίο. Σε σχέση και με τη χρήση. Και αυτοί οι ορισμοί ίσως θα πρέπει να είναι ακριβέστεροι από την αόριστη κατηγοριοποίηση που υπάρχει τώρα. Χρειάζεται πιο συγκεκριμένη προσέγγιση. Έχουμε ετοιμάσει κάποιες ιδέες, να τις συζητήσετε, αν σκεφτείτε. Δεν είναι τόσο βασικές για τη λειτουργία της οδηγία. αλλά η αναθεώρηση της οδηγία για τα σκάφη αναψυχή δεν συμβαίνει πολύ συχνά και σαν νομοθέτε, έχουμε δικαίωμα να, να ρίξουμε ιδέες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν κάποιες ε, λεπτομέρειες που αναφέρω, διότι εξετάσαμε αρκετά ενδελεχώς το θέμα, Κάνετε κάποιες προτάσεις, κάναμε προτάσεις χρήστες διαφόρων κατηγοριών σκαφών, από ναυπηγοβιομηχανίες και από αρχές που είναι υπεύθυνε για τη δοκιμή των σκαφών και τις εποπτικές αρχές. Θέλαμε να διευκολυνθεί η κατάσταση, θέλαμε να βελτιώσουμε την εκνευσιμότητα των σκαφών, κυρίως λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σκάφη είναι σχετικά κινητά αγαθά και ελεύθερα μετακινούνται από χώρα σε χώρα. Θυμάμαι όταν πήγαμε σε μια αποστολή στην περιοχή της, ε, του Φάμπς και της Κέπχαρτ, στη λίμνη Κωνσταντζα και ακούσαμε εξαγωγή σκαφών από την Ελβετία προς Γερμανία που γίνεται σχετικά εύκολα. Ξεκινάει κανείς από την Ελβετία, οδηγεί ε, το σκάφος του στη λίμνη και μετά καταλήγει σε άλλη χώρα. Λοιπόν, θέματα Μετακίνηση είναι πάρα πολύ σημαντικά στον τομέα αυτό των θρασίων μεταφορών. Θέματα ευθυνών για τα εισαγόμενα σκάφη. Χρειάζονται κάποιοι ορισμοί και οι προδιαγραφέ ασφαλεία πρέπει να γίνουν αυστηρότερε για τα σκάφη που έχουν χώρου διαβίωση Εκεί υπάρχουν ανησυχίες για θέματα ηλεκτρισμού, φυσικών αερίων, μόνωσης των ε, δεξαμενών ε, καυσίμων κλπ. που όλα αυτά είναι σημαντικά για την ασφάλεια των θαλασσίων μεταφορών. Και υπέβαλα σχετικά τροπολογίες. Εν γέννη, με τα χαράς ε, σας υποβάλλω την έκθεσή μου προς συζήτηση στην Επιτροπή και χαίρομαι που κάποιοι συγγητές και σχεδόν συγγητές είναι παρόντες. Αυτό προτείνω είναι ε, να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων σχετικά με αυτά που προτείνω και μετά θα καλέσω το Λουί Φιλίπ Ευζηράο που είναι επικεφαλής μονάδας και είναι υπεύθυνος για το θέμα αυτό να εκφράσει από Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις προτάσεις μου και μετά μπορούμε να προχωρήσουμε και να πάμε στο επόμενο στάδιο των τροπολογιών. Ας κάνουμε λοιπόν ένα γύρο συζητήσεων, να σας ακούσουμε απόψεων των συζητητών. Ο κ. Σφάπ είναι εδώ, η κυρία Γκέπχαρτ, ξέρω θα μιλήσει για τον κ. Ρίπερ, ο κ. είναι εδώ, ο κ. Διόν δεν είναι εδώ. Ο κ. Ρούπερ είναι εδώ. Άντριο Σβάμπ, λοιπόν. Α, η κυρία Γκέφχαρτ θα ξεκινήσει. Καλημέρα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Προσωπώ τον σκιώδη εισηγητή της ομάδας μου, κύριο Ρορέπο, που δυστυχώ σήμερα το πρωί θα προσέθει από την Φινλανδία. Δεν έφτασε, αλλά με ειδοποίησε ώστε να το γνωρίζω περί τίνος πρόκειται. Πρέπει να πω ότι το ταξίδι σε σχέση με την ε, λίμνη της Κωνσταντίας ήταν πολύ ενδιαφέρον και ήταν ενδιαφέρον το ότι μπόρεσε να γίνει αυτό και μάλιστα με τόσο μεγάλη ταχύτητα ήταν ένα ωραίο, μια ωραία εμπειρία και φτάσαμε σόι και αυλαβής από πλευράς του συναδέφου χαιρετίζει πολύ το σχέδιο έκθεσης στο οποίο έχει υποβληθεί και το βρίσκει ιδιαίτερα ενδιαφέρον το ότι οι πτυχέ τη ασφάλεια καλύπτονται με ιδιαίτερο τρόπο. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό. Και οι προτάσει ε, και όσα λέγονται για τι εκπομπέ ρήπων και την ε, ηχητική, την ε, ηχητική ρήπανση είναι βιώσιμα πράγματα και θετικό βρίσκει επίσης και την ένταξη των βιοκαυσίμων που ανταποκρίνονται σε σχέση με τον τομέα των αναγκών που υπάρχουν σε σχέση με τα ε, σκάφη υψηλής, υψηλότερης ταχύτητας ε, και επιδόσεων. Οι βελτιώσεις λοιπόν της ε, οριζόντιας, των οριζόντιων ρυθμίσεων πιστοποίησης και των ελέγχων προϊόντων είναι και αυτά σημεία τα οποία είναι σημαντικά και τα χαιρετίζει ο συνάδελφος και αυτά. Και μια και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση 97% βρίσκονται παραγωγή των σκαφών αυτών και είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το βρίσκει ιδιαίτερα σημαντικό ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει με αυτόν τον τρόπο να λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη, διότι είναι ένας τομέας στον οποίο εργάζονται και είναι σημαντικός. Επίσης ο συνάδελφος είναι πεπισμένος ότι συνεισφέρει για την βελτίωση της ασφάλειας των προϊόντων αυτή η προσπάθεια και έτσι θα ενισχυθεί η θέση των καταναλωτών. Να προσθέσω κάτι εδώ υπό το πρίσμα μου, ακριβώς όσον αφορά την ηχητική όχληση, την εκπομπή ε, θορύβων, είναι σωστό ότι δεν αφορά όλους, όλες αυτές τις, ε, όλους τους θορύβους. Όμως κάθε προσπάθεια πρέπει να καταβληθεί ώστε να μειωθεί η ηχητική ρήπανση, γνωρίζοντας ότι οι ιδιοκτήτες αυτών των ε, σκαφών επιδόσεων και υψηλών ταχυτήτων θέλουν να ακούγεται ο θόρυβος της μηχανής τους, ε, όμως παρόλα αυτά πρέπει να υπάρξουν και κάποια όρια. Πιστεύω ότι αυτό το οποίο αναφέρατε σε σχέση με αυτό το θέμα είναι πραγματικά αξιόλογο, διότι ξέρουμε ότι εδώ και το ίδιο, η ίδια η πλεύση των σκαφών στο ε, νερό επηρεάζεται και μπορεί και αυτή η κρούσια ας το των σκαφών στο νερό να συνεισφέρει και αυτή να μειωθεί ο θόρυβος. Θα τα δούμε όλα αυτά. Ευχαριστώ. Ähm, Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς Πρόεδρε ως εισηγητή για αυτή την έκθεση, για αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία για τα αθλητικά σκάφη και να ευχαριστήσω και για τη συνεργασία με τις άλλες ομάδες που ήταν υποδειγματικοί. και μπορούμε να πούμε έτσι ότι είναι πολύ ισορροπημένη η έκθεση και περιεκτική και σκόπιμη. Εγώ πιστεύω ότι η διατήρηση των τιμών ε, για τις εκπομπές ρήπων είναι σωστή για τη βιομηχανία και η ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι το αντιμετωπίζει. Και στο τέλος τέλος έχουμε τις πιο αυστηρές προδιαγραφές παγκόσμια για, αυτές ε, τις, για αυτή την προσέγγιση. Και για τα αθλητικά σκάφη, για τα σκάφη επιδόσεων είναι σωστό να είμαστε φιλόδοξοι και να κάνουμε αυτό το φιλόδοξο βήμα. Είναι ευχάριστο το ότι ίσως θα μπορούσε να υπάρξει μια παγκόσμια ενιοποίηση, τυποποίηση, διότι η παραγωγή τέτοιων σκαφών βρίσκονται και σε άλλες χώρες και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Και από την άλλη πλευρά η κυρία Γκέπχαρτ το προανέφερε, οι τιμές, οι ωριακές τιμές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Από την άλλη πλευρά η μη ρύθμιση ή με την αρχή της επικουρικότητας το να αφήσουμε τους κανόνες αυτούς να διαμορφώνονται από τα κράτη-μέλη, μια και βλέπουμε απλά ότι εδώ υπάρχουν περιφερειακές διαφορές και για την λειτουργία σε μικρέ λίμνες τέτοιων σκαφών υπάρχουν τελείω διαφορετικέ προδιαγραφέ από ό,τι σε με πολλά νησιά για παράδειγμα, σε ανοιχτό πέλαγος. Εδώ λοιπόν πρέπει να υπάρχει κάποια μικρή διαφοροποίηση, ιδιαίτερα όσον αφορά και το κόστο το οποίο θα μπορούσε να εκραγεί και να, εξογω... να διονγκωθεί. Γι' αυτό πρέπει να διαφοροποιούμε τα πράγματα. Το θέμα στη Γερμανία σε σχέση με την εφαρμογή αυτή τη οδηγία όσον αφορά εισαγωγή, ιδιωτική εισαγωγή τέτοιων σκαφών πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, διότι σε σχέση με το γερμανικό δίκαιο, οι εισαγωγέ, οι ιδιωτικές εισαγωγές δεν ενέπιπταν στο πλαίσιο αυτής τη οδηγίας. Πέρα από αυτό υποστηρίζουμε επίσης την εκπόνηση ε, μιας ρύθμισης για νέε κατηγορίες σκαφών ή πλοίων. Έτσι, ένας ολόκληρος τομέας ε, εδώ θα μπορεί να αναφέρεται για την βελτίωση αυτής της οδηγίας και αυτό είναι κάτι πολύ θετικό πιστεύω. Θα με ενδιαφέρε να ακούσω από εσάς κύριε Σίγητα τι γίνεται με την τροποποίηση των κατηγοριών. Είχατε προτείνει, αν τα θυμάμαι σωστά, από την τελευταία συνάντηση σκιοδοτών έχουμε μία νέα επίπτωση μελετών Impact Assessment. Θα με ενδιαφέρε να γνωρίζουμε πού βρισκόμαστε και σε σχέση και με την Επιτροπή. Και αν έγκαιρα πριν από την ψήφιση μπορούμε να τα έχουμε αυτά. Αλλά είμαστε ικανοποιημένοι με την έκθεση μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Uh, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι έξω και δουλειά, Πρόεδρε. Το έχουμε συνηθίσει όμως. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ που σε αυτό το κείμενο. Ε, νομίζω ότι είναι καλό να προσπαθήσουμε να, να, πώς να το πω, το θέμα των εκπομπών, των εξατμίσεων, να το ευθυγραμμίσουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο διαγραφές. Διότι όπως είπε και ο Ανδρέας, εργαζόμεθα σε ένα παγκόσμιο επίπεδο με τα σκάφη και τα ατομικά σκάφη και τα σκάφη αναψυχής και μπορούμε να εισαγάγουμε ε, παγκόσμιες ε, προδιαγραφές για την αυσιπλοεία. Τεχνικά, πολύ καλά. Έδωσε κάποιες πληροφορίες για τις κατηγορίες των σκαφών, σχεδιασμού. Ε, ήθελα να το ζητήσω αυτό, αλλά έδωσε ήδη απάντηση. Χαίρομαι το, ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, λαμβάνονται υπόψη και η θέση τους, διότι τα περισσότερα σκάφη αυτά, τα μικρά, κατασκευάζονται σε μικρό αριθμό από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χαίρομαι επίσης που μέγιστη ηχητική πίεση κυρίως για τα jet έχει μειωθεί γιατί είναι μεγάλο πρόβλημα στα σκάφη αναψυχής. Έχω ερώτηση. Χρειάζεται να είναι υποχρεωτικό τα σκάφη τα οποία έχουν τουαλέτες που είναι αναγκαίες ότι πρέπει να αναφέρονται στην νομοθεσία αυτά τα σκάφη ή να τα αφήσουμε στην αγορά τη ρύθμιση ή να έχουμε υποχρεωτική πρόβλεψη για την απομόνωση των ε, δοχείων των δεξαμενών ύδατος ε, για να μην μολύνουν τα ποτάμια, να υπάρχει μια μόνωση ούτως ώστε να μην μυρίζουν τα ποτάμια από τις τουαλέτες. Και μετά το σήμα ΙΣΥ e ευρωπαϊκή κοινότητα. Χρειάζεται καλύτερος έλεγχος για, ε, για τη χορήγηση αυτού του σήματος. Καλό είναι να χορηγούνται, αλλά πρέπει να ελέγχουμε τη σωστή χορήγηση. Μετά, για ασφαλέστερο και καθαρότερο περιβάλλον, ίσως σαν πρόεδρο θα μπορούσατε να συντάξετε, να στείλετε μια επιστολή μάλλον, προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών, να εισαγάγει μια ευρωπαϊκή άδεια για τα σκάφη. Ήδη είπατε ότι είναι εύκολο να πάει κανείς να περάσει από χώρα σε χώρα και σε μια χώρα είναι κάτι υποχρεωτικό να έχει άδεια για το σκάφος και σε άλλη δεν είναι υποχρεωτικό και να υπάρχει και ισότιμο, ισότιμη όρη στην Ευρώπη για να έχουμε ένα ασφαλέστερο περιβάλλον. Γι' αυτό θα πρέπει να θεσπίσουμε μια βάση όσον αφορά τη χορήγηση αδείας για τα σκάφη αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως πρέπει να μιλήσουμε στον εισηγητή της Επιτροπής Μεταφορών. Ε, μπορεί ενδεχομένως να κάνει παράλληλη δήλωση και ο αρμόδιος ε, επίτροπος. Ε, ενδεχομένως να είναι ο καλύτερος τρόπος να το κάνουμε. Μπορούμε βέβαια να το συζητήσουμε. Η κυρία... Θα με εξέπλητε αν αυτό δεν είχε υποβληθεί ως πρόταση από πλευρά του συναδέλφου. Τυπικό είναι αυτό βέβαια. Όμως και εγώ θέλω να ευχαριστήσω εσάς για αυτή την έκθεση. Έτσι όπως βλέπω εγώ τα πράγματα και όπως τα έχουμε συζητήσει, πολύ λίγες ανάγκες υπάρχουν για τροπολογίες. Ένα σημείο θα ήθελα μόνο να συζητηθεί περισσότερο. Η κυρία Γκέπα το προανέφερε με θετικό τρόπο. Εγώ με αρνητικό τρόπο θα το προσεγγίσω. Το θέμα των βιοκαυσίμων από φυτικά, από φυτά. Υπάρχουν νέε μελέτε που δείχνουν ότι η παραγωγή τέτοιου είδου ε, ε, βιοκαυσίμων από φυτά απαιτεί μεγαλύτερες ποσότητες καυσίμων. Και όλοι γνωρίζουμε το πρόβλημα όσον αφορά την παραγωγή ε, προϊόντων για σύντηση επισητιστικές ανάγκες. Γι' αυτό θα ήθελα να το αφήσουμε αυτό εκτός. Θα ήθελα την υβριδική δυνατότητα κινητήρων να την εξετάσουμε, διότι είναι μια εξέλιξη που είναι πραγματικά σκόπιμο να καλυφθεί και έτσι και σε ε, αυτές τις τροπολογίες θα πρέπει να μπορέσει να καλυφθεί. Πολύ αργότερα σε μια νέα αναθεώρηση θα προχωρήσουμε κατά τα άλλα. Όπως είπα όλα βαίνουν καλώς και όλα είναι εντάξει και για τη στρατηγική σε διεθνείς προδιαγραφές που πρέπει να προσεγγίσουμε και να μην έχουμε ξεχωριστές προδιαγραφές μόνο για την Ευρώπη. Πρέπει φυσικά να μεριμνήσουμε οι εξαγωγικές δυνατότητες για την Ευρώπη να παραμείνουν ανοιχτές. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς άλλος να σχολιάσει. Αν όχι να απαντήσω. Κύριε Γκέπχαρ, θέλετε να κάνετε ένα επιπρόσθετο σχόλιο. Ήθελα στην παρατήρηση της κυρίας Ρούλε να αντιδράσω. Δεν μίλησα για φυτικά βιοκαύσιμα, αλλά μόνο για βιοκαύσιμα. Εντάξει. Και δεν είναι ακριβώς ο ίδιος ο ορισμός. Αυτό ήθελα να παρατηρήσω. Ευχαριστώ. Okay, well, I'll come back on that. Θα επανέλθω σε αυτό Πολύ σύντομα, αν δεν θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο. Αν δεν θέλει κανείς άλλος το λόγο, να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίως για την αναθεώρηση των προτύπων σχεδιασμού, την οποία πρότεινα. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες ε, με επεξηγήσεις στην ε, έκθεσή μου. Νομίζω ότι το σημαντικό είναι ότι δεν είναι κάτι το οποίο μόνοι μας το, αναπτύξαμε, το συζητάμε εδώ και καιρό. Στο πλαίσιο μιας, ε, ενός προτύπου ISO, εναρμονισμένου, ευρωπαϊκού, δεν, ε, είναι μια συζήτηση που δεν την έχουμε ενσωματώσει εδώ, αλλά θα ήθελα να ακούσω την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα αυτό. Αν θεωρούμε ότι είναι σημαντικό αυτό το θέμα, μπορούμε να έχουμε και μία σύντομη έκθεση εμπειρογνωμόνων για το θέμα αυτό. Αλλά θα ήθελα να ακούσω πρώτα τι έχει να πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την έκθεσή σας. Μπορούμε να συμφωνήσουμε με τις περισσότερες τροπολογίες και προτείνουμε να εγκριθούν. Έχουμε κάποιες ανησυχίες όμως στο θέμα των κατηγοριών ε, σχεδιασμού, γιατί αυτή η συζήτηση λαμβάνει χώρα από το 2004. Και στο πλαίσιο της, ε, παρουσία, της ε, προετοιμασίας συγκεκριμένης έκθεσης, η δυνατότητα προσαρμογής και αλλαγής των κατηγοριών συζητήθηκε επίσης. Είναι αρκετά περίπλοκο ζήτημα κατά την άποψή μας και δεν είμαστε σε θέση να συγκεράσουμε τις απόψεις των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών ε, ειδικότερα όσον αφορά τον ενδεχόμενο αντίκτυπο που μπορεί να έχουν ε, οι συγκεκριμένες αλλαγές ε, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οπότε, από τεχνικής απόψεως μπορούμε να κάνουμε τις αλλαγές. Νομίζουμε όμως ότι θα χρειαζόταν μια λεπτομερής μελέτη αξιολόγησης αντικτύπου όχι μόνο όσον αφορά τον αντίκτυπο από οικονομικής και κοινωνικής απόψεως, αλλά και του κατά πόσο, πώς θα τι είδους θα πρέπει να είναι αυτές οι τεχνικές ε, αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Θα ήθελα επίση να πω, σε σχέση με τις τροπολογίες 21 ε, έως 27, θα θέλαμε να διατηρήσουμε όλες αυτούς τους όρους που αναφέρουμε και τους έχουμε αντιστοιχεί συγκεκριμένες κατηγορίες, ε, παράκτια, υπεράκτια, εσωτερική ναυσιπλοεία κλπ. Γιατί θεωρούμε ότι είναι σημαντική πληροφορία, ειδικότερα για το μέσο καταναλωτή. Οπότε, Εντάξει, είναι γεγονό ότι ο αέρα και ε, τα κύματα είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά νομίζουμε ότι είναι σημαντικέ και οι πληροφορίε που ανέφερα. Θα θέλαμε επίση να σε επιστήσουμε την προσοχή στην τροπολογία 32 που αναφορά στο κίνδυνο ανατροπής του σκάφους, γιατί ήδη η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, κάπως ε, πιο ήπια καθιστά της, ε, την νομοθεσία, η οποία αναφέρει ότι κάποια κράτη, κάποια σκάφη, συγγνώμη, δεν έχουν αυτόν τον κίνδυνο, δεν παρουσιάζουν αυτόν τον κίνδυνο. ότι δεν υπάρχει δηλαδή αυτός ο κίνδυνος και γι' αυτό δεν πρέπει να γίνει αξιολόγηση κινδύνου για να φανεί ακριβώς ότι δεν υπάρχει ο κίνδυνος. Αν δεν γίνει όμως αυτή η, κίνδυνη, η κίνδυνη, αν δεν γίνει αυτή η αξιολόγηση κινδύνου, τότε τα πρότυπα πλοημότητας πρέπει να, είναι, να παραμείνουν στα επίπεδα που έχουμε σήμερα. Έχουμε και μερικά λιγότερο σημαντικά ζητήματα βέβαια, τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε διμερώς, αν θέλετε, κυρίως σχόλια διατύπωσης, αλλά κατά βάση αυτά είναι τα δύο βασικά ζητήματα που είναι ιδιαίτερη σημασία για μας. Και βεβαίως Ευχαρίστω να παράσχουμε οποιασδήποτε πληροφορίες σε σχέση με την αξιολόγηση αντικτύπου. Όλα τα δεδομένα, όλες τις πληροφορίες που έχουμε από τις μελέτες ε, που έχουμε εκπονήσει για να διευκολύνουμε τις σχετικές εργασίες. Ευχαριστώ. Uh, well, thank you very much uh, for your Ευχαριστώ πολύ. <laughs> Έχουμε λίγο χρόνο και θα ήθελα να το θέσω το θέμα αυτό. Το θέμα της κατασκευής των ε, σκαφών ε, που έχει να κάνει με πολλές μικρομοσίες επιχειρήσεις, γιατί αυτές είναι κυρίως οι κατασκευάστριες εταιρείε. Επίσης υπονοήσατε κάτι για την αλλαγή στον, κατηγορίε κατηγορίες ε, σχεδιασμού ότι θα ήταν κάπω μειονεκτική η αλλαγή που προτείνουμε για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Μήπω μπορείτε να μα πείτε για ποιο λόγο το πιστεύετε αυτό. Γιατί εμένα με ανησυχεί αυτό και άλλους μπορεί να τους ανησυχεί. Είναι πραγματικά ένας σοβαρός φόβος για την ε, πρόταση, για την έκθεση που ε, έχω συντάξει. Ο εκπρόσωπος Επιτροπής. Δεν ξέρουμε γιατί η αξιολόγηση αντικτύπου δεν έγινε και γι' αυτό δεν ξέρουμε ποιος είναι ο αντίκτυπος. Αλλά είναι γεγονός ότι οι κατηγορίες σχεδιασμού ε, σημαίνουν ε, πιο ε, αυστηρά, αυστηρές προδιαγραφές σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για παράδειγμα, να σας δώσω ένα παράδειγμα για την τροπολογία 22 οι υφιστάμενες διατάξεις επιτρέπουν να τοποθετούνται στην αγορά τα σκάφη αν ε, πληρούν την ε, απέτηση ε, για ισχύ κατηγορία 8 ενώ αυτό που προτείνει τώρα η τροπολογία υπονοεί ότι η ισχύ του ανέμου πρέπει να είναι 10 αντί για 8. Δηλαδή είναι πιο αυστηρή η απέτηση αυτή που τίθεται. Οπότε, το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε και για την τροπολογία 23. Με τη νέα τροπολογία απαιτείται όλα τα σκάφη να συμμορφώνονται τουλάχιστον ε, με ύψος κύματος 7. Δεν ξέρουμε αν η πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μπορούν να συμμορφωθούν με αυτές τις απαιτήσει. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι μια λεπτομερής ε, αξιολόγηση αντικτύπου θα ήταν ευπρόσδεκτη. Αλλά όπω είπα και προηγουμένως, ένα από τα βασικότερα προβλήματα που έχουμε μέχρι τώρα είναι ότι δεν μπορούμε να βρούμε συνένεση μεταξύ των, ενδιαφέρον, των ενδιαφερομένων μερών και των ε, κρατών μελών για το θέμα αυτό. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Πριν συνοψίσω. Μήπως ε, θέλει κανένα συνάδελφος ή σκιώδη εισηγητής ε, να πει κάτι σε σχέση με αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Μάντες. Ναι, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την ευρωπαϊκή άδεια χρήση σκαφών. Δεν ξέρω αν είναι υπεύθυνο γι' αυτό, αλλά μπορεί να έχει, να έχει μια άποψη. Έχετε το λόγο. Κοιτάξτε, εμείς ε, υποστηρίζουμε την ιδέα Γνωρίζουμε τα προβλήματα βέβαια που θα αντιμετωπίσουμε στο Συμβούλιο σε σχέση με τέτοιου είδους διάταξη. Μάλιστα, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μία κρούση στην Επιτροπή Μεταφορών ε, βάσει των όσων είπαμε και προηγουμένως, επειδή ε, εξετάζουμε και τις ανησυχίες των πελατών στην εσωτερική αγορά ε, και νομίζω ότι είναι κάτι που οι ε, πολίτες ε, θα το βρουν ιδιαίτερος ενδιαφέρον, θα τους αρέσει πολύ. Νομίζω ότι μπορούμε να το συζητήσουμε και να το προωθήσουμε. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να συνοψίσω και να σας δώσω και τις σχετικές ημερομηνίε. Από ό,τι κατάλαβα από αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον να συνεχίσουμε με μια πιο λεπτομερή εξέταση των κατηγοριών των σκαφών, να δούμε δηλαδή τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Και θα ζητήσω, αν συμφωνείτε από τη Γραμματεία, να δούμε κατά πόσο μπορεί ένας ε, ειδικό ανάδοχος ε, να αναλάβει αυτή την εργασία και μάλιστα το συντομότερο δυνατόν για να μπορέσουμε να ε, είμαστε εντό του χρονοδιαγράμματό μα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα πρότεινε πρόσβαση και σε περισσότερε πληροφορίε αν, χρειασ... αν, το αν τις χρειαστούμε. Ε, θα το αναλάβω εγώ ως εισηγητής και βέβαια θα ενημερώσω και τους σκιώδεις ε, εισηγητές για τις σχετικές εξελίξεις. Τώρα, για κάποια άλλα λεπτομερέστερα σχόλια για το θέμα των βιοκαυσίμων. Καταλαβαίνω τα ζητήματα που έθεσε η κυρία Ρούλη, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν δύο σημαντικά ζητήματα. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να κατηγοριοποιήσει τα βιοκαύσιμα με πολύ συγκεκριμένο τρόπο ε, και όποια καύσιμα ε, υπάρχουν κάποια καύσιμα που δεν θεωρούνται βιοκαύσιμα και τα οποία δεν ε, εξετάζονται ως τέτοια στην πρόταση. Ούτως ή άλλως υπάρχει μια πρόταση που αφορά τα βιοκαύσιμα και είναι ορισμένα πράγματα που πρέπει να τα λάβουμε υπόψη και για το βιοδίζελ και για τα βιοκαύσιμα όταν ε, μιλάμε ε, για τις εκπομπές των σκαφών. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι καλύπτονται αυτά τα πράγματα βέβαια είναι γεγονός ότι δεν είναι πάντοτε τα καύσιμα που χρησιμοποιούν ε, τέτοιου είδου καύσιμα. Βέβαια, στο Βορρά, στη Σουηδία για παράδειγμα, βιοκαύσιμα χρησιμοποιούνται σε σκάφη αναψυχή σε μεγάλο βαθμό δεν είναι θέμα αύξηση ή μείωση χρήση βιοκαυσίμων, είναι θέμα πρακτικό. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι ε, μηχανέ των σκαφών ε, έχουν ε, την κατάλληλη επίδοση και να προσπαθήσουμε να, να επιτύχουμε έναν στόχο εκπομπών αερίων όποιου είδους καύσιμα και να χρησιμοποιεί το σκάφος. Για τα άλλα γενικά ζητήματα, οι συνάδελφοι από ό,τι κατάλαβα είναι ικανοποιημένοι. Αν όμως έχετε και άλλες ιδέες και ειδικότερα για ζητήματα που έχουν να κάνουν με μικρότερους κατασκευαστές ε, σκαφών, ε, να εξασφαλίσουμε δηλαδή να, να, να, το ότι δεν θα είναι τεράστιες οι απαιτήσει, ε, να εξασφαλίζονται κάποιες απαιτήσει περιβαλλοντικές και δημόσιας ασφάλειας, είναι γεγονός ότι πολλές φορές κάποιοι αγοράζουν ένα σκάφος και στη συνέχεια το τροποποιούν και πρέπει να εξασφαλίζουμε ότι δεν θα το αποθαρρύνουμε αυτό. Πρέπει κάποιος να καταλαβαίνει μεν τι θα πει από άποψη κατασκευής ε, σκάφους ε, μια καλή πρακτική και ενδεχομένως μάλιστα να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα σε κατηγορίες καφών που ούτω ή άλλω είναι επιστοποιημένα. Όσον αφορά τώρα τα, το χρονοδιάγραμμα, μισό λεπτό να βρω τα χαρτιά μου. Τροπολογίες μέχρι τις 27 Μαρτίου, 12 το μεσημέρι. Στην Επιτροπή Μεταφορών και Περιβάλλοντος ε, θα ψηφίσουμε 24-25 ε, του Απρίλη και εμείς τότε θα εξετάσουμε τις δικές μας τροπολογίες για να περάσει στην Ολομέλεια της, ε, του Μαΐου. Εν τω μεταξύ ελπίζουμε να μπορέσουμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα που έχουμε με τις κατηγορίες σχεδιασμού που αναφέραμε προηγουμένως για να μπορέσουμε να λάβουμε και τις πληροφορίες αυτές υπόψη. Μέχρι τις 27 Μαρτίου λοιπόν υποβολή τροπολογιών, αλλά θα κάνουμε και μια συνάντηση σκιωδών εισηγητών νωρίτερα. Ευχαριστούμε πολύ. Να έχουμε προχωρήσει λίγο πιο γρήγορα το προβλεπόμενο, διότι θα έχουμε μια παρουσίαση μια εκθέσεω που αναθέσαμε ε, με βάση κάποιες τροποβολογίε που πρότεινε η Επιτροπή και χρειαζόμαστε τον εισηγητή και άλλους. Η κυρία Βέσφαλ είναι εδώ, έχουμε έναν βασικό σκιώδη εισηγητή. Προτείνω το εξή. Σύντομο διάλειμμα. Δεκάλεπτο. Θα αρχίσουμε ακριβώς στις 9.55 με παρουσίαση από τους εμπειρογνώμονες και συζήτηση για τις συνέπειες που έχουν οι τροπολογίες που προτείναμε. Θα ξαναρχίσουμε ακριβώς στις 9.55. Ευχαριστώ. για Ο κύριος Βαντεκάμπαρ είναι, ξανά, είναι εδώ μαζί μας, οπότε ξαναρχίσουμε συνεδρίαση. Θα ασχοληθεί λοιπόν ε, με το επόμενο θέμα. Θα ήθελα την προσοχή σας, σας παρακαλώ, Τουάν Τουάν Μάντερς. Τουάν Τζιμ είναι ο λόγος. Νομίζω ότι όλοι οι σκιώδες είναι παρόντες για τη συζήτησή μας. Περαιτέρω συζήτηση όσον αφορά το στάδιο που, στο οποίο βρισκόμαστε για την οδηγία για τα μοτοποδήλατα και να συζητήσουμε όμως περισσότερο αυτό που ζητήσαμε, την αξιολόγηση συνεπιών. Ε, με βάση τις τροπολογίες που υποβάλαμε. Γιατί ζητάμε σημαντικές αλλαγές προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία που έχουμε συνάψει με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκεί που προτείνουμε σημαντικές αλλαγές, λέγει ότι θα πρέπει να ζητήσουμε κάποια εξωτερική συμβουλή και ανάλυση των συνεπειών που έχουν αυτές οι αλλαγές όσον αφορά το τελικό αποτέλεσμα και το κόστος πρότασης. Και νομίζω ότι παίρνει σοβαρά αυτή την ευθύνη η Επιτροπή μας και το αποδεικνύει η πρότασή μας. Είναι η πρώτη φορά σε αυτό το κύκλο εργασιών της Επιτροπής όπου καλέσαμε να διεξαχθεί μια ανάλυση από πλευρά συμβούλων και να έρθουν σύμβουλοι και να παρουσιάσουν τα συμπεράσματά τους. Και οι σκιώδεις εισηγητές που πρότειναν τις αλλαγές θα υποβάλουν ερωτήσεις. Αυτό θα κάνουμε όταν γίνει η παρουσίαση της μελέτης και μετά οι σκιώδεις εισηγητέ θα παρουσιάσουν ερωτήσεις και θα ακούσουμε και τι έχει να πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε τον Φιλίπ Τιζού και την ομάδα του από το τμήμα των οχημάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε τον κύριο Βανταϊκάπ που είναι υπεύθυνο για το όλο εγχείρημα και θα κάνει με σύντομη εισαγωγή και μετά θα δώσω στον κύριο Μόρις Γκουτέλ από το London Economics ε, θα κάνει παρουσίαση και ο κύριος Πάτρικ Μούρες από την London Economics ο κ. Βάνταν ο εισηγητή, θα κάνει μια εισαγωγή. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι σωστό είναι από πλευρά ε, του London School of Economics πρώτα να ακούσουμε τι απόψει του σχετικά. Γνωρίζω ότι οι συνάδελφοι αυτή την έκθεση σίγουρα διεξοδικά θα την έχουν μελετήσει και εξετάσει. Υπάρχουν αρκετά θέματα που πρέπει να συζητηθούν. Λογικό όμω είναι πρώτα να ακούσουμε την πρόταση, μετά τα σχόλια. Okay, well, well, let's do that. Καλώς, αυτό θα κάνουμε. Ακούστηκε ότι είσαστε London School of Economics, αντί η εταιρεία σας λέγεται London Economics, έτσι. Εντυπωσιάστηκα τόσο πολύ από το London School of Economics, τα μπέρδεψα, ξέρετε. London Economics, το έκανα London School of Economics. Λοιπόν, εσεί κύριε και έχουμε και τι διαφάνειε και έχουμε και αντίγραφα των διαφανειών και όλοι έχουν αντίγραφα των διαφανειών και τι εκθέσει, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ναι, καταρχά την πρώτη διαφάνεια γίνεται μια επισκόπηση των όσων θα αναφέρω. Θα κάνω μια σύντομη εισαγωγή περιγράφοντας κάποιες κοινέ υποθέσεις επί των οποίων βασιζόμεθα και μετά θα αναφερθώ σε συγκεκριμένους τομείς στους οποίους αναφέρεται η αξιολόγηση αντικτύπου και μετά θα ακολουθεί συζήτηση. Αν πάμε στο όλο ιστορικό, πρόκειται περί των συνεπειών. Βάση είναι διάφορες τροπολογίες που υπευλήθησαν στην πρώτη ευρωπαϊκή Επιτροπής για κανονισμούς για τα οντομέτων μοτοποδηλάτων. Πιο συγκεκριμένα, καλύπτει Τρει τομεί αυτή η αξιολόγηση συνεπειών. Οι αυξημένε απαιτήσει για την ασφάλεια, ABS και σύστημα τροχοπέδησης που δεν μπλοκάρουν οι πτωχοί, μετά τα συστήματα διάγνωσης στο όχημα και αλλαγή χρονοδιαγράμματος για την εφαρμογή σε μεταγενέστερο στάδιο των προδιαγραφών περί εκπομπών καυσαερίων. Πήραμε την πρόταση σαν βάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξετάσαμε τις αλλαγές που εισάγονται μέσω των τροπολογιών. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπουμε τι κάναμε, την προσέγγιση. Πήραμε την αξιολόγηση συνεπειών που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή ήταν η αφετηρία μας. Και για τα ποιοτικά μας συμπεράσματα χρησιμοποίησαμε λίγο πολύ αυτή τη βάση και αναφερθήκαμε και στις πηγές που χρησιμοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Νοσολογικής Συνεπιών και τις δύο εκθέσεις με το εργαστήριο έρευνας και την έκθεση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Πήγαμε και σε, κάναμε διαβουλεύσεις με τους βασικούς εμπλεκομένους φορείς. Δεν έγινε πλήρης διαβούλευσης. Συνομιλήσαμε με εκπροσώπους του τομέα, των μοτοποδηλάτων, των κατασκευαστών, κάποιους κατασκευαστές, Honda, Triumph, λάβαμε γραπτά σχόλια. Μιλήσαμε με την Ένωση Μοτο... Χρήστων Μοτοποδηλωτών και τον έλεγχο μέσω καταλητών των εκπομπών. Ήρθαμε σε επαφή με διάφορους εκπροσώπους δηλαδή. Στην επόμενη διαφάνεια αναφέρομαι σε κάποιες κοινέ υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν στην αξιολόγηση αντιχτύπου. Προσπαθήσαμε στο βαθμό του δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε κοινέ υποθέσεις για να είναι τα αποτελέσματα σύνεπη, όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και κάποιες υποθέσεις όσον αφορά τον πληθωρισμό, όπως σε πρώτερες έρευνες. κάναμε διαχωρισμό μεταξύ νέων τύπων και υφισταμένων τύπων στην καταχώρηση οχημάτων. Είναι σημαντικό για τα ποσοτικά αποτελέσματα αυτός, ο διαχωρισμός είναι σημαντικός. Και τις παρούσες τιμές μέχρι το 2021, 2012-2021. Τιμές καταναλωτού για τα μοτοποδήλατα. Βασιστήκαμε στα πιο καλά 50 μοντέλα σε κατηγορία από, από πρώτη θέση μέχρι πεντηκοστή. Βασικές διαφορές με την πρώτερη δουλειά ήταν επικαιροποίηση των προβλέψεων για νέες καταχωρήσεις. Αν δείτε τον πίνακα αριστερά, το γράφημα, αυτές είναι οι προβολές που χρησιμοποιήθηκαν το 2009 που τονίζονται, βασίζονται στα πορίσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, μελέτη αντικτύπου. Χρησιμοποίησαμε επικαιροποιημένα ε, στοιχεία για τις νέες ε, καταχωρήσεις. Βασικά χρησιμοποίησαμε το ίδιο μοντέλο, το χρησιμοποίησαν οι ίδιοι άνθρωποι με πιο σύγχρονα στοιχεία όμως. Μετά εξετάσαμε συγκεκριμένα τα πρώτα μέτρα για τις απαιτήσει ασφαλείας, τις βελτιωμένες απαιτήσει ασφαλείας. Αυτή η διαφάνεια δείχνει το status quo της Πρωτάς Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποχρεωτικό ABS για βαριές μοτοσυκλέτες από το 2017 και υποχρεωτικό ABS ή e CPS ή και τα δύο για ελαφρότερες μηχανές. Η πρώτη αλλαγή είναι η εισαγωγή του ABS ένα χρόνο νωρίτερα. Επόμενη αλλαγή. Ε, επέκταση των απαιτήσεων σε εφιστάμενα οχήματα. Άλλη αλλαγή για τις ελαφρές μοτοσυκλέτες, επέκταση της απέτηση για ABS αντί CBS σε αυτή την κατηγορία των οχημάτων. Εντοπίσαμε τις βασικές συνέπειες όσον αφορά τις αξιολογήσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είδαμε το κόστος κατασκευής, πώς επηρεάζεται και εκτιμήσαμε και την αποφυγή ατυχημάτων από την πλευρά ωφελών άλλες υποθέσεις που έγιναν 30-70 χωρίσαμε βαριές μοτοσυκλέτες από πιο ελαφριές μοτοσυκλέτες 500 ευρώ αναόχημα για το ABS το μισό κόστος 250 ευρώ για CBS συνδυασμένο σύστημα τροχοπέδησης και ίσως αυτό θα επανέλθουμε στο κόστος. Γιατί αμφισβητούνται. Οι προμηθευτές θεωρούν ότι ίσως το κόστος να είναι το 1 πέμπτο αυτού του υπολογισμένου ποσού, ίσως 100 ευρώ. Άλλες υποθέσεις. Αποτελεσματικότητα των συστημάτων πέδησης από μια έκθεση που έχει διεξαχθεί από ευρύτερη έρευνα που είχε διεξαχθεί. Είναι ευρύ θέμα αυτό. Εμείς πήραμε ως βάση τους αριθμούς σαν δεδομένα. Υπολογίσαμε τους θανάτους, θανάσιμα ατυχήματα ανεόχημα όχημα για τα διάφορα είδη μοτοσυκλετών και συστημάτων τροχοπέδησης. Τέλος. Κάναμε μια αξιολόγηση τραυματισμών και θανάτων που απεφεύθησαν. Κοινό τρόπο αυτό αξιολόγηση, έχουμε διάφορα στοιχεία. Χρησιμοποίησαμε αυτά που χρησιμοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αξιολόγηση συνεπειών. Βάσει όλων αυτών των υποθέσεων, έχουμε ποσοτικά αποτελέσματα για το κόστος και το όφελο για τις δύο κατηγορίες οχημάτων, βαρύτερες κατηγορίες Α2 και Α3 και ελαφρύτερες μοτοσυκλέτες κατηγορία Α1 βλέπουμε ότι το κόστος του μέτρου εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα του ABS όπως είδαμε, δηλαδή πόσοι θάνατοι απεφεύθησαν. Περισσότεροι αποφεύγονται με τη χρήση του ABS. Και η θνησιμότητα, ένα ποσοστό θνησιμότητας μετεβλήθη σε σοβαρούς τραυματισμούς. 747 εκατομμύρια, 1,2 δις κόστος για τα βαρύτερα οχήματα, 95% αυτού οφείλεται στην επέκταση των μέτρων στα ισοσυσίοντες τύπους, 383 θάνατοι αποφεύγονται με τη χρήση του EBS. Αυτό είναι το όφελος. Άρα οικονομίες 380 εκατομμύρια. Ελαφρύτερα οχήματα. Α1. 610 εκατομμύρια με 761 εκατομμύρια όσον αφορά το κόστος. 96% οφείλεται στην επέκταση των μέτρων στα εφιστάμενος τύπους οχημάτων. Ξέρουμε για τις ελαφρύτερες μοτοσυκλέτες που είναι φθηνότερες. Η αύξηση του κόστους που θα είναι αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ABS είναι αρκετά σημαντικό ποσοστό του συνολικού κόστους. Έχει 18%. Η εισαγωγή όμως το EBS αποφεύγει, οδηγεί στην αποφυγή 155 θανάτων. Άρα εξοικονομούμε ένα εκατομμύριο αναθάνατο. Άρα εξοικονομούμε 153 εκατομμύρια. Αν τα προσθέσουμε όλα αυτά, το καθαρό κόστος του μέτρου είναι 1,4 δις. Αν υποθέσουμε υψηλότερη αποτελεσματικότητα εμπειρίας, πάμε στο 1,9 δις. Αν δεν είναι τόσο αποτελεσματικότητα εμπειρίας. Με βάλαμε, μετά είδαμε τι γίνεται αν προσθέσουμε συστήματα διαγνωστικά στο όχημα. Βασιστήκαμε στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή είναι η βάση. Υποχρεωτική χρήση. Του σταδίου 1 για μοτοποδήλατα και μοτοσικλέτες για το 2017. Και το 2021 ξεκινάει η δεύτερη φάση. Οι τροπολογίες προβλέπουν εισαγωγή για το OBD1 και OBD2 ε, ένα χρόνο νωρίτερα για μοτοσικλέτες κατηγορίας 3 να μπουν αυτά τα συστήματα τα διάγνωση Και επέκταση του συστήματος στα ήδη υπάρχοντα οχήματα, σε υπάρχουσες κατηγορίες για τα μοτοποδήλατα, εισάγεται η απέτηση για τη χρήση στι υπάρχουσες κατηγορίες αλλά η απέτηση για να εφαρμοστεί το δεύτερο στάδιο των συστημάτων διάγνωσης αφαιρείται, υπάρχει μόνο τη κατηγορία 1. Όσον αφορά τι συνέπειε, εντοπίσαμε το κόστο του να μπει ο εξοπλισμός βασικό στοιχείο του κόστους και η μείωση εκπομπών, στόχος που είναι του μέτρου αυτός, που είναι όφελος. Υπάρχουν και άλλα ωφέλη. Πολύ μικρά, σε κάποιες περιπτώσεις, ή δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν. Κάναμε και άλλες υποθέσεις για να υπολογίσουμε το κόστος όφελος. Υποθέσαμε ότι το διαγνωστικό σύστημα 1 είναι βασικό προϊόν, 11 ευρώ ανά όχημα είναι το κόστος, είναι απλό προϊόν, βάσει στοιχείων που έχουμε από το Ηνωμένο Βασίλειο, από το Υπουργείο Μεταφορών του Ηνωμένου Βασιλείου. Το κόστος της δεύτερου σταδίου του διαγνωστικού συστήματος είναι 46 ευρώ ανά όχημα. Εμείς ακολουθήσαμε συντηρητική προσέγγιση από τα στοιχεία που διατίθενται. Δείχνουμε τι σημαίνουν τα στοιχεία στο εδώ όσον αφορά ποσοστό λιανικής τιμής του οχήματος. Χρησιμοποιώντας αυτές τις υποθέσεις που ανέφερα, υπολογίζουμε το συμπληρωματικό κόστος το καθαρό 130 εκατομμύρια ευρώ για αυτό το μέτρο. Και όπως και πριν, βασικός οδηγός είναι η επέκταση του μέτρου στα υφιστάμενα ίδιο οχημάτων. Εύκολο να το καταλάβετε αυτό. Γιατί. Διότι οι υφιστάμενοι τύποι είναι πολύ μεγαλύτερο κομμάτι του συνολικού νέου στόλου, του συνολικού στόλου, 80% κάθε χρόνο. Στη διαφάνεια Βλέπετε το διαχωρισμό των αποτελεσμάτων κατά κατηγορίες οχημάτων. Είδαμε πώς μειώνονται οι εκπομπές. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι αλλαγές λόγω τροπολογιών θα ήταν ελάχιστες στον φάρτης εκπομπές. Δεν φαίνονται στο γράφημα. Εάν βάλει τα στοιχεία στη γραφική παράσταση. Τελευταίο μέτρο χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των προδιαγραφών για τι εκπομπέ. Αρχική πρώτη Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν το Euro 3 για νέους τύπους από το 2014 και για υφιστάμενους τύπους το 2015 και μετά 2017-2018 Euro 4 και 2020-2021 το επόμενο στάδιο, για υφιστάμενου τύπους. Η τροπολογία ΣΥΜΚΟ προτείνουν το βήμα γύρω 3 να φύγει. και ταχύτερη εισαγωγή του σταδίου γύρω 4 για το 2016 για νέα, οι νέους τύπους και 2017 για εφιστάμενους τύπους. Εξετάσαμε το περιβαλλοντικό κόστος. Τα στοιχεία μας δείχνουν ότι θα είναι ελάχιστο. Η μείωση εκπομπών ανά είναι αρκετά σημαντική, σύμφωνα με τις απαιτήσεις Euro 4. αλλά δεν, λόγω της τροποποίησης δεν αλλάζουν πάρα πολλοί εκπομπές, λόγω της ήδη επιτυχανόμενης μείωσης, λόγω των προτάσεων Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γενικά υπάρχουν πιο αυστηρές απαιτήσεις που οδηγούν σε περισσότερη καινοτομία στη τεχνολογία των κινητήρων και αυτό ίσως οδηγήσει στο ότι θα γίνει πιο ανταγωνιστική ευρωπαϊκή βιομηχανία. Αυτό αμφισβητείται όμω από του κατασκευαστέ. Αυτό ήταν το θεώρημα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λένε ότι υπάρχουν υψηλοί δασμοί κατασκευαστέ. Και ίσω οι εξαγωγέ να μην είναι, πάνε τόσο καλά. Δεν το λάβαμε αυτό υπόψη. Ε, δεν κάναμε ποσοτικοποίηση αυτών των στοιχείων. Δεν τα λάβαμε υπόψη αυτά. Εκτιμήσει κόστο για το βήμα Euro 4. Καθορίζει την έκθεση LAT, αυτή που χρησιμοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το κόστος θεωρείται από κάποιους ότι είναι, θα είναι πραγματικά τετραπλάσιο από αυτό που υπολογίζουμε εμείς που είναι 50 ευρώ. Δηλαδή να φτάσει μέχρι 200 ευρώ. Ανάλογα με τις υποθέσεις που ακολουθεί κανείς, Ίσως τελικά έχουμε σημαντική αύξηση της λιανικής τιμής της μοτοσυκλέτας. Κυρίως αν πάτε να δείτε την κατηγορία των μοτοποδηλάτων, που είναι τα φθηνότερα οχήματα. Πήραμε νέα στοιχεία. Πόσα οχήματα ήδη συμμορφώνονται με τα νέα όρια εκπομπών που προτείνονται από την ΙΜΚΟ. Πήραμε στοιχεία από τη Γερμανία. Το 1 τέταρτο περίπου των νέων οχημάτων πληρούν τις νέες προδιαγραφές. Αυτό δεν συμπεριλαμβάνει όμως τα κριτήρια βιωσιμότητας, διαρκείας των οχημάτων και αντοχής τους. Δεν ποσοτικοποίησαμε ακριβώς τι γίνεται ανάλογα με τη χρήση του οχήματος και τη φθορά του και τα χιλιόμετρα που είχε κάνει. Θεωρήσαμε ότι 25% των οχημάτων ήδη συμμορφώνονται με τις νέες διαγραφές. 50 ευρώ αν όχημα κοστίζει αυτό. Υπολογίσαμε. Με βάση αυτό έχουμε συμπληρωματικό κόστος 16 εκατομμύρια ευρώ θα μπορούσε να είναι και ψηλότερο κόστο. Περιβαλλοντικό όφελο. Μικρό. Αυτά βρήκαμε στην αξιολόγηση συνεπειών. Σα ευχαριστούμε πολύ, πολύ καλά. Σε σχέση με τα πολύ χρήσιμα στοιχεία, σε σχέση με τα, διαγρα... με τα γραφήματα, να ελπίζω ότι το κείμενο θα μπορέσει να είναι στη διάθεση όλων για να υποφεληθούν όλοι. Αυτό που θα κάνω τώρα θα είναι θα προσκαλέσω να ακούσουμε τα σχόλια των σχεδόν εισηγητών. Κάποιες ερωτήσεις και σε εσά επίσης. Και έτσι ίσως θα μπορούσαμε να καλέσουμε τον εισηγητή ο ίδιος να παρέμβει γιατί γνωρίζει περισσότερα από τους άλλους. Ιδιαίτερα όμως να μας πει αν θεωρεί ότι η μελέτη επιπτώσεων, impact assessment, θα έπρεπε να οδηγήσει σε κάποιες αλλαγές σε σχέση με την τοποθέτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά και τα μέλη της ίδιας μας Επιτροπής. Ε, και θα καλέσω τους άλλους σκιώδεις εισηγητές, την κυρία Βέσφα, τον κύριο Μάντας, την κυρία Ρούλα και, τα, και Και εγώ ίσω θα μπορούσα να σχολιάσω στο τέλο. Ο κύριο Φάντερ πρώτο παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω ότι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησα τα της μελέτης επιπτώσεων που αναφέρθηκαν. Και στην εισαγωγή ήδη αναφέρθηκε. Επομιζόμαστε τις ευθύνε μας με ιδιαίτερα σοβαρό τρόπο και με μεγάλη χαρά συνεργάστηκα ώστε να μπορέσουμε αυτή τη μελέτη επιπτώσεων να την ζητήσουμε να μας υποβληθεί. Θα ήθελα να πω ότι μας δίνει κάποια περισσότερα στοιχεία σε αυτά που θέλουμε να πετύχουμε και στο έργο που θέλουμε να επιτελέσουμε. Να επενθυμίσω κάτι σύντομα, ότι όλη αυτή η, όλος αυτός ο κανονισμός συντάσσεται από πλευράς μας για να έχουμε μια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή βιομηχανία όσον αφορά τα δίκυκλα αυτά ή τα οχήματα, στα αποκαλέσουμε έτσι αυτά, που θα πρέπει να είναι καλής ποιότητας ε, η παραγωγή μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Θα μπορούν έτσι λοιπόν να προσαρμοστούν. Θα πρέπει να είναι ασφαλής αυτή η παραγωγή και καθαρή όσον αφορά το περιβάλλον. Φοβούμαι ότι η μελέτη επιπτώσεων όσον αφορά αυτούς τους στόχους ε, δεν μπορεί να παραμείνει χωρίς κάποιες επικρίσεις. Τα αποτελέσματα πιστεύω δεν δίνουν λύσεις για τις συζητήσεις και τα ζητήματα που ανεφίσαν κατά τις συζητήσεις μας. Μια και είναι πιο περιπλόκα και πιο σύνθετα κάπως τα πράγματα από ότι ανέφεραν οι ερευνητές ή εξέτασαν και καταδεικνύουν οι ερευνητές στις μελέτες τους. Θα αναφερθώ σε αυτά. Η πρώτη επίκριση λοιπόν είναι και εκείνη από το σημείο με ποιον συζήτησε κανείς και τι έγινε δεκτό. Και σε σχέση με τους επένους που μπορούν να γίνουν δεκτοί για αυτές τις παρατηρήσεις και το συνεπαγόμενο κόστος που το αναφέρουν οι μελετητές. Λένε θα υπάρξει ένα τέτοιο κόστος. Όμως το κόστος των 500 ευρώ το οποίο ήδη είναι υψηλό και θα αυξάνεται ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Αυτό είναι κάτι λοιπόν το οποίο πρέπει να το λάβουμε έτσι υπόψη και να το κρίνουμε αντικειμενικά σε αυτό το πλαίσιο. Δεύτερο, η ε, Net Present Value uh, μέθοδος, NPV, μέθοδος δηλαδή που καταδεικνύει το καθαρό, την καθαρή ε, ενισχύ αυτή τη στιγμή πρόσθετη αξία. Και πρέπει εδώ να πούμε ότι βλέπουμε το NPV να αναφέρεται και να λαμβάνεται υπόψη να δεν καλύπτει όλες τις πτυχές αυτής της μελέτης. Το ABS για παράδειγμα όσον αφορά τα ελαφρότερα οχήματα για παράδειγμα τα μοτοποδήλατα. Και αυτό δημιουργεί κάποια σύγχυση σε σχέση με νέους τύπους και ήδη υφιστάμενους τύπους και στους πίνακες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διαφοροποιούν σε σχέση με υποχρεώσεις, σε σχέση με τα σημερινά ενισχύει ε, για τα οχήματα αυτά και για τα νέα και τις νέες υποχρεώσεις. Αυτή η διαφοροποίηση δεν είναι πάντα σαφής ε, στην έκθεση των πραγματογνωμόνων. Τουλάχιστον αυτό πιστεύω εγώ και έχουμε και για την μεθοδολογική προσέγγιση των ατυχημάτων είναι νομίζω θα έλεγα από πλευράς των αριθμητικών αυτών μεγεθών για τις ε, βαριές μεγάλες κατηγορίες και για τις ε, ελαφρότερες κατηγορίες είναι αριθμητικά μεγέθη που πρέπει να λάβουμε ιδιαίτερα υπόψη ως πολιτική στην πολιτική μας ευθύνη και για το OBD2 ε, το on diagnostics 2, το κόστος το οποίο θα συνεπάγεται αυτή η προσέγγιση πρέπει να ληφθεί υπόψη, να τα σταθμίσουμε με την συνολική κατάσταση αυτά τα κόστη και νομίζω ότι θα είναι υπεύθυνο να εισαχθεί το, ε, η προσέγγιση αυτή. Το ίδιο λοιπόν ε, ισχύει και για τις ε, προδιαγραφές για τις εκπομπές ρήπων. Με ικανοποίησε όταν άκουσα να αναφέρεται ότι για τον, τους παγκόσμιους, στην παγκόσμια σκηνή ανταγωνιστές μας πρέπει να ισχύουν αυτά. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία είναι πολύ καλή και έχει καλές επιδόσεις. Όταν τέτοια θα ισχύουν τώρα, τέτοιες απαιτήσει θα ισχύουν, να λάβουμε υπόψη την Κίνα, την Ινδονησία, που με τέτοιου είδους μοτοποδήλατα και ε, μοτοσυκλέτες δημιουργούν πολύ μεγάλα προβλήματα στην ρήπανση του περιβάλλοντος και το κόστος το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη και αυτό πρέπει να ε, είναι νομίζω ε, κάτι το θετικό. Μία συγκεκριμένη ερώτηση τώρα. Για αυτή τη μελέτη και για τις προτάσεις που μας υποβάλλετε σε σχέση και με το ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο και την ε, Επιτροπή ΙΜΚΟ θα έπρεπε να αλλάξουν, να τροποποιηθούν όλα αυτά. Θα λέγα όχι ως απάντηση, όχι σε αυτή τη φάση. Οι αριθμοί, τα αριθμητικά μεγέθη είναι θα έλεγα αμφίσιμα. Δεν μπορεί κανείς μόνο σε αυτά να βασίζεται. Θα πρέπει με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσουμε προς ποια κατεύθυνση μπορεί να βρεθεί μια λύση. Είχαμε τον τελευταίο καιρό πολλές άτυπες συναντήσεις και υπό τη Δανέζικη Προεδρία που γνωρίζουμε ότι είναι πρόθυμη να προβεί σε συμβιβασμούς είναι σημαντικό με τη γνώση αυτή των μελετών επιπτώσεων να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτές τις άτυπες συζητήσεις. Ευχαριστώ. Η κυρία Βέστφα. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρωτού τώρα πω κάτι περισσότερο για αυτή τη μελέτη. Θα ήθελα να πω κάτι σε σχέση με την ψηφοφορία για εντολή για την πρώτη ανάγνωση. Επιβεβαιώνω για άλλη μια φορά εδώ ρητά και κατηγορηματικά για τη δική μου κοινοβουλευτική ομάδα ότι εξακολουθούμε να ενδιαφερόμαστε με το ίδιο αυτό πρότυπο όπως και με την έκθεση Πανσέρι να προβούμε στον τριμερή διάλογο. Αναμένω ότι ο εισηγητής τώρα γοργά θα προχωρήσει στην εκτέλεση αυτής της εντολής, θα πάρει αυτή την εντολή και θα προχωρήσει στις διαπραγματεύσεις για λογαριασμό μας. Τώρα, να επισέλθω στη μελέτη του London Economics. Έχω κάποιες ερωτήσεις για τους συντάκτες αυτής της μελέτης. Πρώτη ερώτηση. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος παράγει αυτά τα ABS, τα συστήματα μη, ε, του, να μην μπλοκάρουν τα, φρέμα, τα, τα φρένα. Είναι η παραγωγή των ε, ε, εξαρτημάτων ή κάποια άλλη παραγωγή θα έλεγα όταν γνωρίζουμε και θέλουμε να μάθουμε το κόστος για ένα τέτοιο εξοπλισμό ABS θα ζητήσουμε αυτή την πληροφορία από τον ίδιο τον παραγωγό, από εκείνους που παράγουν τα εξαρτήματα μεμονωμένα ή και τους δύο. Η μόνη βάση δεδομένων που ε, αναφέρετε εσείς είναι εκείνη του, ε, του, της Ένωσης των Παραγωγών. Όμως από τους ίδιους τους παραγωγούς εξαρτημάτων δεν βλέπουμε να υπάρχουν κάποια στοιχεία. Εσείς ισχυρίζεστε στη σελίδα 10 της μελέτης ότι ρωτήσατε λέει αυτούς τους παραγωγούς ε, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Ένωση Παραγωγών, ούτε ένας από αυτούς δεν ρωτήθηκε από εσά, ούτε ήρθατε σε επαφή ούτε και με έναν από αυτούς. Πώς επεξηγείτε αυτό. Τι έχετε να πείτε. Επιπλέον δημιουργείται το ερώτημα για μένα. Πώς μπορεί να αξιολογήσει κανείς το κόστος κάποιου πράγματος χωρίς να είχε ερωτηθεί ο υπεύθυνο εκείνος που παράγει τις συσκευές ή τον εξοπλισμό. Λέτε 500 ευρώ είναι το κόστος ρεαλιστικά εξεταζόμενο για το ABS. Την πραγματική τιμή πώλησης για μια Yamaha XJ για παράδειγμα μπορείτε να μας την αναφέρετε αυτή είναι 500 ευρώ σε σχέση με τους καταναλωτές νέου είναι κάτι λιγότερο από 500 όμω ευρώ, πράγματι θα έλεγα. Η τιμή αγοράς τώρα για τους παραγωγούς όσον αφορά την κάλυψη των εξαρτημάτων από τους παραγωγούς εξαρτημάτων και ανταλλακτικών είναι 120 ευρώ περίπου. Και κάτι ακόμα το οποίο πρόσεξα σε σχέση με τη μελέτη σας. Λέτε και κινείται από το στοιχείο ότι μόλις το EBS λέτε το 17 θα ε, ισχύει υποχρεωτικά για όλους, το κόστος ανά ABS μονάδα θα αυξηθεί, λέτε. Αυτό μου φαίνεται πραγματικά να είναι κάτι μοναδικό και ανεπανάληπτο, ασύλληπτο στην ιστορία της βιομηχανίας οχημάτων και δικύκλων. Κύριε Χάβερ, εσείς ο ίδιος προέρχεστε από την αυτοκίνητο βιομηχανία. Σίγουρα θα συμφωνήσουμε ότι η θέση και η τοποθέτηση ότι κάθε εμπειρία και κάθε βίωμα σε σχέση με αυτού του είδους θέσεις α, αντιφάσκει. Γιατί να είναι επιπλέον α, δαπανηρότερο για τους παραγωγούς όταν θα είναι υποχρεωτικό για όλους. Και γιατί ετήσια αυτό το κόστος να συνεχίσει να αυξάνεται. Παρακαλώ να μου απαντήσετε αυτό το ερώτημα εδώ και τώρα. Παράλληλα με αυτά τα οποία αναφέρετε υπάρχουν πολλά σημεία στη μελέτη για μένα που πραγματικά με κάνουν να δυσανασχετώ και να μην μπορώ να τα δεχτώ και στο τέλος θα ήθελα να τονίσω κάτι. Πώς εσείς αντιμετωπίζετε αυτά τα στοιχεία και πώς μας παρουσιάζετε αυτά τα αριθμητικά στοιχεία. Τα στοιχεία της SM τα είχαμε πριν από ένα χρόνο στη διάθεσή μας. Επίσης το ίδιο και την μελέτη της TRR, Transport Research Laboratory και της Επιτροπής. Πιστεύετε κυρίες και κύριοι ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καταλήγουμε σε συμπεράσματα. Ευχαριστώ. Κύριε παρακαλώ. Σα ε, Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ προσθέτω τη φωνή μου στις απόψεις των προλαλισάντων. Όμως, θα ήθελα να πω ότι η έκθεση είναι θετική, πιστεύω. Έχει θετικά στοιχεία, διότι μας κάνει να ανοίξουμε τα μάτια και να μας πούν ότι βρισκόμαστε στη σωστή πορεία και κατεύθυνση. Είμαστε στο παρελθόν και εξακολουθούμε να είμαστε στη σωστή πορεία και κατεύθυνση. Και γιατί. Διότι πιστεύω ότι οικονομικά εμείς η Ευρώπη ως η πλουσιότερη, η πιο ευημερούσα Ήπειρος πρέπει να έχουμε ρόλο προπομπού και πρωτοπόρων όταν θέλουμε να παράγονται ασφαλείς κινητήρες και οχήματα. Το ίδιο είπαμε και για τα σκάφη πιο πριν. Πρέπει να είμαστε εμείς ε, η αιχμοί του δόρατος, η προπομπή, οι πρωτοπόροι και για τις προδιαγραφές που θα εισαγάγουμε θα πρέπει να προσπαθούμε να διαχέονται παγκόσμια ώστε να γίνονται αποδεκτές παντού. Όταν έχουμε και τους παραγωγούς της ίδιας της Ευρώπης που σε σχέση με τα όσα παράγουν στην ε, ε, ευρωπαϊκή αγορά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι αυστηρότατες προδιαγραφές οι οποίες πολλές φορές είναι και επώδυνες. Όμως είδαμε ότι στην έκθεση σε σχέση με τις θέσεις απασχόλησης μπορεί να μην δημιουργούνται τόσες πολλές περισσότερες θέσεις απασχόλησης αλλά όμως δεν μειώνονται και θέσεις απασχόλησης. Τουλάχιστον πρέπει να είμαστε προς μια σωστή πορεία. Και ένα άλλο θέμα. 380 εκατομμύρια λέει επιπλέον κόστος θα δημιουργηθεί, αν τα θυμάμαι καλά τώρα, πάμπολες ζωές, ανθρώπινες ζωές μπορούν να διασωθούν και φυσικά όταν θέλουμε να, και μπορούμε να σώσουμε αυτές τις ζωές ε, με σχετικά μικρές επενδύσεις, αξίζει σίγουρα η προσπάθεια και ο κόπος. Αυτή η πορεία που υιοθετήσαμε και ακολουθούμε είναι λοιπόν η σωστή. Και μπορεί κανείς να πει ότι μπορεί ίσως να έχει κάποια αρνητή, κάποιες αρνητικές πτυχές αυτή η έκθεση, όμως μας δείχνει ότι βρισκόμαστε στη σωστή κατεύθυνση και γι' αυτό είμαστε ευγνώμονες, γιατί μπορούμε να δούμε ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Με ικανοποιεί λοιπόν αυτή η έκθεση. Και να κάνω και μια άλλη παρατήρηση όσον αφορά την πλευρά εισηγητού. Την έκθεση αυτή θέλαμε, θέλαμε να δημιουργήσουμε μεγαλύτερο πλαίσιο ασφάλειας, μεγαλύτερη ασφάλεια. Κάποια θέματα ίσως δεν έγιναν δεκτά, όμως θα πρέπει να δούμε ότι σε σχέση με τον ε, κανονισμό αυτά τα πράγματα που εντάχθηκαν πρέπει να προχωρήσουν Είμαι ευγνώμων λοιπόν γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ε, Η κυρία Ρούλε, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θέλω ακριβώ να συνεχίσω από αυτό το οποίο είπε ο κύριο Μάντα, όταν είπε ότι είναι ικανοποιημένο με αυτή την έκθεση. Εγώ μπορώ να πω ότι δεν είμαι ικανοποιημένη με αυτή την ανάλυση. Δεν πιστεύω ότι μα βοηθάει να κάνουμε ούτε ένα βήμα προ τα εμπρό. Το αντίθετο, οπισθοχωρούμε μάλλον. Και θέλω να διατυπώσω το ερώτημα, Πώς δίνουμε εντολή για τέτοιες αναλύσεις, διότι κοστίζουν κόστος και δαπάνες ε, για το Κοινοβούλιο. Αναμένω από τέτοιες αναλύσεις ευθύ εκ προημίου να καθίσταται σαφές ότι εδώ έχουμε κάποιο πρόβλημα, τριβές αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα μεταξύ παραγωγών και το οχημάτων και παραγωγών ανταλλακτικών ε, και εξοπλισμών πρέπει να δούμε ότι θα πρέπει να ανατρέχουμε και στα αριθμητικά μεγέθη αμφωτέρων. Εδώ δεν έγινε όμως αυτό. Πρέπει να γίνεται. Ένα άλλο τμήμα όπου περιμένω να υπάρχει μεγαλύτερη ενιοποίηση είναι το κόστος μεταξύ ε, πώλησης ε, και κέρδους. Πρέπει να δούμε ποιο είναι το περιθώριο κέρδους, ιδιαίτερα όταν αφορά τον μη υποχρεωτικό εξοπλισμό. Το ίδιο πρόβλημα είχαμε και με καταλήτες και με διάφορα άλλα μέσα και εξοπλισμούς και συσκευές. Στην αρχή τα περιέγραψαν όλοι πανάκριβα. Στη συνέχεια όμως όταν έγιναν υποχρεωτικά μειώθηκαν οι τιμές τους όταν έγινε υποχρεωτικός αυτός ο εξοπλισμός. Θέλω όλα αυτά λοιπόν να αναλυθούν σε σχέση με τις υποχρεώσεις των παραγωγών και σε σχέση με τη διαμόρφωση του κόστους, ώστε να έχουμε μια καλή βάση για σύγκριση. Δυστυχώς δεν έγινε όμως αυτό. Το τελευταίο σημείο. Θα ήθελα και πρέπει να πω ότι ανέμενα το κόστος των εκπομπών ρήπων και το κόστος των ατυχημάτων και το κόστος των ε, ανθρώπινων ζωών που χάνονται ως θύματα από τέτοια ατυχήματα. Όλα αυτά να λαμβάνονται υπόψη και να καλύπτονται σε σχέση με τα συστήματα ABS για παράδειγμα. Uh, uh, Ευχαριστώ. Ένα σχόλιο από δική μου πλευρά για ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα. Η βασική μου ανησυχία για την ανάλυση του ABS είναι για τα μικρότερα οχήματα, όπου υπήρχε μία πρόταση να έχουμε ένα συνδυασμένο σύστημα τροχοπαίδηση, ε, το οποίο θα είναι φθηνότερο και απλούστερο από το ABS. Και από ό,τι κατάλαβα, υπήρξε και ένα συγκεκριμένο πίνακα που μα παρουσιάσετε από αυτού, που επιβεβαιώνει τι δικέ μου απόψει ότι υπάρχει μια διαφορά ε, κόστους και απλότητας ε, για τα μικρότερα, μικρότερης απόδοσης ε, οχήματα σε σχέση με τα μεγαλύτερα. Ίσως θα μπορούσατε να το σχολιάσετε, αλλά σε γενικές γραμμές συμφωνώ με τα σχόλια των συναδέλφων. Δεν ξέρω αν η κυρία Ρόιτοβα θέλει να πάρει το λόγο, αλλά θέλει και ο πρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής να πάρει το λόγο για να μας εξηγήσει ορισμένα πράγματα. Κυρία Γκέπχαρτ, επίσης θέλετε να πάρετε το λόγο. Παρακαλώ, λίγο σύντομα, κυρία Ροϊτόβα, για να έχουμε χρόνο και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομη, γιατί η κυρία Ρούλα τα πεόλα. Με απασχολεί το γεγονός ότι δεν έχουμε αξιολόγηση αντικτύπου της ε, υγείας των θυμάτων, ε, των δυστυχημάτων και δεν είμαι πάρα πολύ βέβαιη για την ορθότητα της προσέγγισης αυτής για τέτοιου είδους ε, οχήματα. Θα έπρεπε να επιτρέπουμε στα κράτη-μέλη να κάνουν κάποιους διαχωρισμούς για να μπορούν κάποια οχήματα να κυκλοφορούν και σε μία χώρα αλλά και σε μία άλλη. Θα ήθελα να ρωτήσω και τον εισηγητή. Τα μοτοποδήλατα, ας πούμε, πώς πιστεύετε ότι μπορούν να ενσωματωθούν στην όλη προσπάθεια που κάνουμε. Ναι, αλλά δεν καλύπτεται από, την, ε, από, τις, ε, από τη συγκεκριμένη νομοθεσία. Άρα τα κράτη-μέλη πρέπει μόνοι τους, μόνα τους να προβούν στις απαραίτητες ε, αλλαγές. Η κυρία Γκέπατ, ευχαριστώ πρόεδρε, θα είμαι σύντομη από πλευρά μου και εγώ. Και να πω ότι σε σχέση με όσα αναφέρθηκαν με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθήσαμε. Δεν έχω ομολογώ ασχοληθεί με αυτό το θέμα και ούτε μελέτησα αυτή τη μελέτη προηγούμενα. Όμως ακούμε εδώ από τον εισηγητή και από σχεδόν, σχεδόν όλους τους σκιώδεις εισηγητές να υπάρχουν επικρίσεις, πολλές επικρίσεις όσον αφορά την ποιότητα αυτής της impact assessment, της μελέτης επιπτώσεων. Νομίζω είναι σοβαρές οι επικρίσεις αυτές και πρέπει να τις λάβουμε σοβαρά υπόψη όλοι. Είναι χρήματα φορολογουμένων εδώ που δαπανούμε των Ευρωπαίων πολιτών. Το οφείλουμε στους Ευρωπαίους πολίτες να μπορούμε να λογοδοτήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο θα πανώνται τα κονδύλια. Και γι' αυτό πρέπει, πιστεύω, το απόγευμα, όταν θα έχουμε τη συνάντηση συντονιστών, να προσθέσουμε ένα επιπλέον σημείο στην ημερήσια διάταξη για, τα, για τις, ε, την ε, ανάληψη της σύνταξης μελετών, τέτοιων μελετών επιπτώσεων. Πώς γίνεται η διαδικασία, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε τέτοιες επικρίσεις εις βάρος τέτοιων μελετών. Και δεν είμαι πρόθυμη εγώ και διατεθειμένη πραγματικά να λένε ότι το Κοινοβούλιο δεν δαπανά σωστά τα χρήματα των φορολογουμένων. Ευχαριστώ. Okay, well, I'm sure that... Uh, Μάλιστα. Ε, φυσικά. Θα το συζητήσουμε και το απόγευμα. Ο κύριος Ντεζόν. Ευχαριστώ πολύ. Δύο σχόλια θα ήθελα να κάνω. Πρώτον για τη διαδικασία και δεύτερον για την περι... περιεχόμενο της έκθεσης. Για τη διαδικασία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ιδιαίτερο το γεγονός ε, ότι, η Ευρω... ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να κάνει αξιολογήσεις ε, των συμβαστικών τροπολογιών, ε, να εξετάσει τα ενδεχόμενο κόστος, όπως επίσης ε, και τον αντίκτυπο των τροπολογιών, ειδικότερα όταν κινούνται προς διαφορετική κατεύθυνση από την αξιολόγηση αντικτύπου που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αρχική της έκθεση. Οπότε, συμφωνούμε με, με την προσπάθεια αυτή σε σχέση με την πρωτοβουλία, ε, και πιστεύουμε ότι είναι ένα συν σε σχέση με την ποιότητα της ε, κοινοτικής ε, νομοθεσίας. Για μας η έκθεση είναι μια έκθεση η οποία συμπεριλαμβάνει κάποια στοιχεία, στοιχεία τα οποία είναι ενημερωτικά. Είναι όμως δύσκολα για μας να πούμε ότι έχουμε στην έκθεση όλα τα στοιχεία που μπορούμε να μας επιτρέψουν να αξιολογήσουμε ε, ε, όλο το, το κόστος και την αποτελεσματικότητα όλων των μέτρων. Δηλαδή βλέπουμε κάποια στοιχεία, αλλά δεν μπορούμε να θεωρήσουμε για τα τρία αυτά θέματα, ας πούμε, ότι έχουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να κάνουμε μία συμπληρωματική αξιολόγηση ε, σε σχέση με αυτή που είχε γίνει από τις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλα στοιχεία, όπως για παράδειγμα στοιχεία τιμολόγησης, κόστους και άλλες μεταβλητές, ε, όπως για παράδειγμα το OBD. Το OBD είναι ένας μηχανισμός που δεν αφορά μόνο περιβαλλοντικές επιδόσεις, αλλά και την αποδοτικότητα της ε, επισκευής, όπως επίσης και τη δυνατότητα των επισκευαστών να μπορούν να παρέμβουν. Υπάρχουν λοιπόν πολλά στοιχεία τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση. Και γι' αυτό διαπιστώνουμε ότι είναι ενδιαφέρουσα η έκθεση, δίνει κάποια στοιχεία, αλλά τα στοιχεία αυτά δεν είναι αρκετά πλήρη για να μπορούμε να κάνουμε μια αξιολόγηση πλήρη. Κατά τη γνώμη μα όμω, ε, σε σχέση τουλάχιστον με τι προτάσει που έγιναν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Um, now, we don't have a lot of time, but I think... Uh, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, αλλά για να είμαι δίκαιο, πρέπει να δώσω στη London Economics τη δυνατότητα να απαντήσει. Γιατί θα κάνουμε και συζήτηση στο μέλλον για αυτό. Μήπω θέλετε να μα απαντήσετε. Και μετά ο κύριο Βαντενκάμπ θα πάρει το λόγο, εισηγητή. I... Ναι. Κοιτάξτε. Πρώτα να πω σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής της μελέτης. Ε, πάρα πολύ στενό για τον αντίκτυπο της υποχρεωτικής εισαγωγής, για παράδειγμα, νέων εξοπλισμών, ε, η εξέλιξη των τιμών, ε, ε, το κόστος της μείωσης των εκπομπών. και τα αποτέλεσμα του συνέπειες του ABS για λιγότερο σοβαρούς τραυματισμούς, για παράδειγμα. δεν είχαμε και πάρα πολύ χρόνο και επομένως και τα αποτελέσματά μας είναι πολύ περιορισμένα. Όσον αφορά τώρα το κόστος ε, για το ABS, που είπαμε ότι είναι 500 ευρώ, ναι, δεν μιλήσαμε με τους κατασκευαστές μεν, αλλά γνωρίζαμε τις εκτιμήσεις κόστους τους και αναφέρονται και στην έκθεση. 500 ευρώ εμένα μου φαίνεται ένα από τα ισχυρότερα ε, νούμερα που αναφέρουμε γιατί βασιστήκαμε στις τιμές, ε, στις διαφορές τιμών ε, μεταξύ μοντέλων που έχουν ABS και μοντέλων που δεν έχουν ABS. Επίσης είμαστε συνεπείς και στο πλαίσιο της έκθεσης γιατί για διάφορα άλλα, για, για άλλο κόστος όπως για παράδειγμα αυστηρότερες προδιαγραφές εκπομπών, OBD και λοιπά χρησιμοποιούμε πολύ πιο συντηρητικά, συντηρητικές εκτιμήσεις. Μας, μας επέκριναν και οι κατασκευαστές. Τα 500 ευρώ λοιπόν, τα 500 ευρώ, λοιπόν ε, βρίσκονται στο πλαίσιο της έκθεσης. Ε, ε, κάποιοι ε, είναι γεγονός ότι υπάρχει, υπάρχουν εκτιμήσεις από 329 έως 800 ευρώ. Εμείς πιστεύουμε ότι το 500 είναι ένας, μια, μια, ένα λογικό νούμερο και μας δίνει μια ιδέα του πώς θα είναι τα πράγματα όταν θα αρχίσει να υπάρχει μια ε, μεγαλύτερος τεχνολογικός εξοπλισμός. Υποθέτουμε ότι θα αυξηθούν και οι τιμές επειδή υπάρχει πληθωρισμός 2% ετησίως. Αυτή είναι μια κοινή πρακτική και τι λάβαμε υπόψη. Έτσι είχε γίνει και στο παρελθόν σε άλλες σχετικές εκθέσεις στον τομέα αυτό. Αυτά ήθελα να πω. Okay. Okay. Um, Mr. Van Ευχαριστώ κύριε Βαντεκάμπ. Σας αφήνω να συνοψίσετε. Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να κινηθούμε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το συμπέρασμα το οποίο μπορώ να συναγάγω είναι ότι η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των μελών αυτής της κοινοβουλευτικής μας επιτροπής θεωρεί ότι επιβεβαιώνονται οι τοποθετήσεις και οι θέσεις μας με τις τροπολογίες ε, που έχουν κατατεθεί. Λέμε και, βλέπουμε ότι πορευόμαστε προς την ορθή κατεύθυνση και πορεία. Εσείς ο ίδιος ε, αναφερθήκατε σε σχέση με τα ελαφρά μοτοποδήλατα και τα λοιπά, το τι πρέπει να γίνεται και πρέπει αυτά να τα λάβουμε υπόψη. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξουμε την κατεύθυνσή μα τώρα. Πρέπει να παραμείνουμε πιστοί στην πορεία που έχουμε υιοθετήσει και θα πρέπει να ψηφίσουμε, να εγκρίνουμε μια εντολή ώστε να μπορούμε να προβούμε σε διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μπορέσουμε να συντονιστούμε για καλύτερου συμβιβασμού μαζί του. Είναι η καλύτερη προσέγγιση, πιστεύω αυτή. Κάθε ένα από εμά και οι συνεργάτε μα καταβάλουμε προσπάθειε και ιδιαίτερε προσπάθειε όλα για αυτό το χαρτοφυλάκιο. Και πρέπει μέχρι την 1η Ιουνίου, ώστε αφορά το Συμβούλιο, να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Αυτή θα ήταν η πρότασή μου λοιπόν. Αύριο θα ήθελα να έχουμε μια σαφή εντολή ώστε να μπορέσω με τους σκιώδεις συζητητές να προχωρήσουμε με τη σωστή αυτή πορεία ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα. Με καλή συνεργασία να καλύψουμε αυτό το χατοφυλάκι όσον αφορά την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Um, Νομίζω ότι αν συμφωνούν οι συντονιστέ, δυστυχώ η κυρία Γκέπχαρτ έφυγε, αλλά φαντάζομαι η κυρία Βέστφαλ συμφωνεί ότι πρέπει να ψηφίσουμε αύριο. Γι' αυτό κύριε Σφαμπ, εσεί τι λέτε. Εντάξει, γνέφει ο κύριο Σφαμπ. Ωραία. Τότε, αν όλοι συμφωνούν, Κυρία Ρούλα, ο κύριος Μάντερς δεν είναι εδώ, οπότε να ψηφίσουμε για την εντολή διαπραγματεύσεων στην αρχή της ψηφοφορίας ε, αύριο, γιατί ξέρετε ότι πρέπει ε, πάνω από τα μισά ε, ε, μέλη πρέπει να είναι εδώ. Ναι, δεν θα ξανακάνουμε το λάθος ε, αυτό, κύριε Κάρμπου, ο κύριος Φαντρικάμπ. Αύριο, λοιπόν, το πρωί, πρώτο θέμα στην ψηφοφορία θα είναι η έναρξη των διαπραγματεύσεων. Κοιτάξτε, ένας από τους στόχους του να έχουμε μια μελέτη αξιολόγησης ε, είναι βέβαια ως ε, εσείς επικεφαλής των διαπραγματεύσεων να μπορείτε να μιλάτε εξ ονόματος της Επιτροπής και Υπάρχουν πάρα πολλές επιπλέον πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για να υποστηρίξετε την άποψη της ε, Επιτροπής μας και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι σημαντικό να υπάρξει ε, μία ακόμη μελέτη. Φαντάζομαι τώρα το πώς θα γίνει αυτό θα το συζητήσετε και με την κυρία Γκέπχαρτ και με τους υπόλοιπους. Γιατί είναι πραγματικά μια πρακτική την οποία θα εξακολουθήσουμε να ακολουθούμε, γιατί ούτως ή άλλως έχουμε τις διαδικασίες μελέτης αξιολόγησης αντικτύπου, αλλά επίσης ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη τις απόψεις όλες των, ε, όλων των ενδιαφερομένων μερών. Ευχαριστώ τη London Economics και όπως είπα θα πράξουμε, αύριο το πρωί θα ψηφίσουμε για τις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ πολύ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία και εκείνη θα συμμετέχει βέβαια στις σχετικές διαπραγματεύσεις. Uh, second, uh, Περνάμε λοιπόν σε μια δεύτερη μελέτη, άλλη μελέτη που ζήτησε η Επιτροπή μας και που πραγματεύεται το θέμα, την εφαρμογή του εξυγχρονισμένου τελωνιακού κώδικα. Από χρωμική απόψεως, είναι πολύ έγκαιρη Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η μελέτη αυτή για τις περαιτέρω εργασίες μας. Ο κύριος Εμέτα θα έρθει σε 11.30 όπως είπα. Μπορεί να συζητήσουμε μαζί του και αυτό το θέμα, να του κάνουμε ερωτήσεις και σχετικά. Νομίζω ότι οι συντάκτες της μελέτης είναι εδώ, από την Price PricewaterhouseCoopers του Βελγίου και της Ολλανδίας. Κύριος Βεστάτε, κύριος Μεζόν, Έτς, Μπρέινε και Μπούβατς. Όλοι εδώ είναι. Είναι όλη η ομάδα των εμπειρογνωμόνων εδώ. Νομίζω η κυρία Λατζέρν θα μιλήσει πρώτη. Η κυρία Λεγκρίπ θα έρθει, είναι η συγκητριά μα, αλλά είναι στην Επιτροπή Εξωτερικών για την ώρα και θα έρθουν και οι σκιώδει εισηγητέ, φαντάζομαι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω εδώ είναι και εκείνη. Καλώ ήρθατε στην ομάδα των τελωνίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αν θέλουν βεβαίω να σχολιάσουν, ευχαρίστω. Πρώτα όμω η κυρία Λατζόιν. Σα δίνω το λόγο, η κυρία Λατζόιν. Έχουμε και διαφάνειε. Εσεί έχετε και αντίγραφα στο φακελό σας. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι τιμή για μένα που είμαι εδώ να παρουσιάσω με μελέτη που ετοιμάσαμε για την Επιτροπή σας όσον αφορά την εφαρμογή του εξεχωρισμένου τελωνιακού κώδικα. Αμέσως θα περάσω στην τρίτη διαφάνεια διότι ήδη έχει γίνει μια παρουσίαση πολύ καλή της ομάδας. Θέλαμε καταρχάς να σας δώσουμε το ιστορικό της σημασίας που έχουν τα τελωνία. Θα εστιαστούμε μεταξύ, μετά στην, στο πεδίο εφαρμογή και μεθοδολογίας μελέτης, τη συλλογή στοιχείων, τα αποτελέσματα αυτής, τι συστάσεις κάνουμε, ποιες είναι ελάχιστες απαιτήσει και ποιο είναι ο κατάλογος επιθυμητών σημείων για τη μελλοντική εργασία. Ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα εξετάζοντας τη σημασία που έχουν τα τελωνία η μελέτη ασχολείται με την εφαρμογή του εξυγχρονισμένου του κώδικα, αλλά αυτό που σίγουρα δείχνει τη σημασία των τελωνίων και γιατί η δουλειά που κάνουμε επί του θέματος ε, είναι σχετική ε, και έχει σημασία. 27 τελωνιακές αρχές υπάρχουν, εποπτεύουν το διεθνές εμπόριο και την ενιαία αγορά. Αυτό, η ενιαία αγορά είναι πιο σημαντική ενότητα εμπορική στον κόσμο, 13.000 δις ευρώ, 13 ευρώ το 2009 αντιπροσωπεύει. Οι τελωνιακέ αρχέ συνέλεξαν αυτό που θεωρούσαμε παραδοσιακού ιδίου πόρου τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, 15% του γενικού προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και ο προπολογισμό του 2012 είναι 19 δις ευρώ. Οι Τελωνιακέ αρχές επίσης Παληθεύουν και ξακριβώνουν περίπου 200.000 ε, ε, διασαφηνίσεις το χρόνο. Και οι τελωνιακές αρχές ε, εμπλέκονται σε μόνιμη διαδικασία εξυγχρονισμού. Εξυγχρονισμός είναι e-customs και συγχρονισμός μέσω λογισμικού όλων των διασαφήσεων και των συναλλαγών ε, και βλέπετε ότι εντό τη προτάσει Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πρόγραμμα ε, βλέπουμε ότι πολλά ε, σημαντικά κονδύλια δίνουν στα τελωνία και μετά θα επιστρέψουμε σε συγκεκριμένο σημείο αργότερα. Σήμερα οι τελωνιακές αρχές λειτουργούν μέσω 27 εθνικών συστημάτων λογισμικού και κάθε χειριστής ε, θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με τα εθνικά συστήματα υπολογιστών του κράτους μέλους του. Αν λειτουργεί σε πάνω από ένα κράτος μέλος, θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με πολλαπλά συστήματα υπολογιστών ε, του κράτων μελών, του κράτους μέλους μάλλον. Μετά θα δώσω στον Dick Hart το λόγο ε, για να σας δείξει τι πεδίο κάλυψε μελέτη και τι, ποια είναι τα υπόλοιπα στοιχεία που καλύψαμε. Ευχαριστώ είναι. Στις 20 Ιουνίου του 2011 ξεκίνησε η μελέτη για να αξιολογήσουμε τις προκλήσεις και τους όρους για την εφαρμογή του εξυγχρονισμένου τελωνιακού κώδικα. Τελειώσαμε τι εργασίε την περασμένη εβδομάδα, την ίδια μέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποθέτησε τον εξυγχρονισμένο κώδικα, τον τελωνιακό. Ο εξυγχρονισμένος κώδικας θα πρέπει να εφαρμοστεί μέχρι 24 Ιουνίου 2013 και γι' αυτό θα έπρεπε καταρχάς να δούμε κατά πόσο αυτή η ημερομηνία μπορεί να τηρηθεί ακόμα, να εντοπίσουμε μεταξύ των βλεκομένων μερών τα ενδεχόμενα προβλήματα, νομικά, τεχνικά και επιχειρησιακά, που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την έγκαιρη εφαρμογή των μέτρων. Και τρίτον, θέλαμε να δώσουμε έναν κατάλογο, τεχνικού προσανατολισμού για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κατάλογο σημαντικών σημείων και του όρου υπό του οποίου θα μπορούσε να εφαρμοστεί ξεχρονισμό του Ελληνικού Κώδικα. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί η μελέτη βασίζεται επί τεσσάρων φάσεων. Η μελέτη εδράζεται επί μελέτη εγγραφών και συλλογή στοιχείων μέσω διαβουλεύσεων με του εμπλεκομένου φορεί. Οι εμπλεκόμενοι φορεί ε, ήταν το Ελεκτικό Συνέδριο, Παϊκή Επιτροπή, 8 τελωνιακέ αρχέ κρατών μελών, 5 ε, οργανώσεις και 16 διάφοροι φορεί σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Μετά αξιολογήσαμε τις προκλήσεις και τους όρους για την εφαρμογή του εξυγχρονισμένου τελωνιακού κώδικα. Από την όλη αξιολόγηση καταλήξαμε σε κάποιες συστάσεις. Μεταξύ άλλων, υποχρέωση να συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των μέτρων. Πρώτη φάση συμπεριλάμβανε την ανάπτυξη του πλαισίου αξιολογήσεω και των διαφόρων ερωτηματολογίων. Δεύτερη φάση. Τα πορίσματα από τη συλλογή των στοιχείων. Πάμε μέσω στη διαφάνεια με τα πορίσματά μας. Πρώτο έβριμα, θέλετε το πόρισμα, ότι ο εξυγχρονισμό του ελληνιακού κώδικα και τις νομοθεσίες θεωρείται πολύ σημαντικός από τον όλο εμπορικό τομέα. Μετά, και, κεντρική διαχείριση τελωνιακή χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να επεκταθεί στα ειδικού φόρου κατανάλωση και το ΦΠΑ, για να ωφεληθεί το εμπόριο. Αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι οι προσπάθειες για ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα πρέπει να συντονιστούν Μία εφαρμογή κατά στάδια ε, δείχνει ότι έχει κάποιες αντιστάσεις στο διάγραμμα. Γιατί υπάρχουν φόβοι ότι θα λειτουργούν διαφορετικά συστήματα και διαδικασίες παράλληλα. Πολλά από τα βασικά πορίσματα έχουν συμπεριληφθεί σε συστάσεις, όπως αυτές που στη διαφάνεια τι χρειάζεται για να υπάρχει σαφή στρατηγική και εναρμόνιση των συστημάτων πληροφορική και πώ μπορούν τα συστήματα να επικοινωνούν καλύτερα μεταξύ του για να διευκολυνθεί το εμπόριο. Κεντρική προσέγγιση για τη χρήση τη τεχνολογία, όπω cloud computing και εμπορικέ έτοιμε εφαρμογέ, είναι κάτι που πρέπει να αξιολογηθεί. Κάναμε διαβούλευση με χώρε. Είδαμε ότι κάποια κράτη-μέλη είναι ανοιχτά να αντικαταστήσουν τεχνικά συστήματα με κεντρικά συστήματα. Άλλα κράτη-μέλη θέλουν να κρατήσουν εθνικά του συστήματα. Κεντρική ανάπτυξη και εθνική ένταξη συστημάτων και ολοκλήρωση μπορεί να γίνει, να το εξεταστεί σαν ενδεχόμενο. Μόνο δύο κράτη-μέλη ήταν κατά αυτή τη ιδέα. 95% του εμπορίου που εξέφασε την άποψή του προτιμά μια κεντρική προσέγγιση όσον αφορά τα συστήματα, τα τεχνολογικά τη πληροφορική. Επιχειρησιακή εφαρμογή του εξυγχρονισμένου τελωνιακού κώδικα αποτελείται από κατάρτιση ανθρώπων και παροχή έγκαιρων και επαρκών πληροφοριών. Οι περισσότεροι εκπρόσωποι του τομέα του εμπορίου πιστεύουν ότι δεν πληροφορούνται επαρκώς. Στην τρίτη φάση, αξιολογούμε τα πορίσματα και θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες στη μελέτη μας. Τέλος, τέταρτη φάση. Εκεί έχουμε τις συστάσεις μας. Γενική σύσταση. Τη βλέπετε στο στοιχείο αυτό. Τέσσερις διαδικασίες που πρέπει να καλύπτονται μέσω ενός ολοκληρωμένου εξυγχρονισμού του ελληνικού κώδικα. Η νομική εφαρμογή, η διαδικασία είναι στο πορτοκαλί χρώμα. Εξυγχρονισμός του ελληνικού κώδικα, η πρόταση για την αναδιατύπωση, έγκριση αυτής, έγκριση των εφαρμοστικών διατάξεων και των καταξιωσιοδότηση πράξεων και θέσπιση εθνικής ομοθεσίας. Κίτρινο τεχνική εφαρμογή. Η διαδικασία θα πρέπει να ξεκινήσει με σημαντικέ αποφάσει για τη στρατηγική πληροφορική. Για το πώ θα κινηθούμε την επόμενη δεκαετία. Θα ακολουθήσουμε κεντρική ή αποκεντρωμένη προσέγγιση για τα συστήματα πληροφορική. Άμα ληφθούν αυτέ οι αποφάσει, χρειάζεται σχέδιο δράση που θα μπορεί να συνταχθεί, να εκτελεστεί και να μεταφραστεί σε εθνικά συστήματα πληροφορικής και τα συστήματα πληροφορική των οικονομικών φορέων. Για να είμαστε σίγουροι ότι γίνεται ομοιόμορφη εφαρμογή τη τελωνιακή νομοθεσία, χρειάζονται προσανατολισμοί για του τελωνιακού και τον τομέα και θα πρέπει να οργανωθεί και η κατάλληλη κατάρτιση. Με το μοβ χρώμα βλέπετε αυτή τη διαδικασία. Τέλο. Το βαθύ κόκκινο δείχνει, το, το πορφυρό χρώμα δείχνει πώ θα ενημερώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα εξασφαλίζεται έτσι η αυστηρή εφαρμογή του γενικού ολοκληρωμένου εξυγχρονισμένου τελωνιακού κώδικα και των συναφών σχεδίων δράσης. Επί τη βάση των πληροφοριών που πήραμε, η βαθμολόγηση με κάποια διευρωπαϊκά δίκτυα, είδαμε ότι στην καλύτερη περίπτωση χρειάζεται 5 χρόνια για εφαρμοστεί το σύστημα. Αλλά μπορεί να φτάσουμε και στα 21 χρόνια. Αυτή είναι η χειρότερη περίπτωση. Συνάδελφός μου, Ρουτ, θα σας καθοδηγήσει στις τελευταίες δύο διαφάνειες. Ευχαριστώ, Ντέρεκ. Αυτά με οδηγούν σε λιγότερα, λιγότερες απαιτήσει ε, για τη διαδοχική εφαρμογή θα δείτε διάφορες παρατηρήσεις για τα 10 αυτά σημεία. Πρώτον, η αναδιατύπωση που δημοσιεύτηκε. εμείς πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνει μια μελέτη εξολόγηση αντικτύπου. Περισσότερες λεπτομέρειες χρειάζονται όσον αφορά την εφαρμογή κυρίω ε, Η αναδιατύπωση αυτή τη στιγμή αφήνει αρκετά πράγματα εκκρεμή. Δύο συστάσεις ε, που βλέπετε στη συγκεκριμένη διαφάνεια αφορούν τη φάση μετά την εφαρμογή. Πρώτο πιστεύουμε ότι το ελεγκτικό συνέδριο πρέπει να υποβάλει έκθεση όσον αφορά την ε, επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα του κώδικα. Και δεύτερον, ε, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τη φάση της, τη φάση εφαρμογής κάθε δύο χρόνια. Ε, στη συνέχεια, σε μεταγενέστερο στάδιο, θα έπρεπε να γίνεται ετησίως. Αν λοιπόν... Ε, δούμε τις ε, απαιτήσεις που υπάρχουν σε δύο διαφορετικά σύνολα. Βλέπουμε την πλευρά της πληροφορικής. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν έκτη, ε, ε, ε, οκτώ συγκεκριμένες συστάσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με τη στρατηγική της πληροφορικής που αφορά αξιολόγηση που πρέπει να γίνει, μια σειρά αξιολογήσεων, μελέτη εφικτότητας για μια προσέγγιση αποκεντρωμένη ή κεντρική, κάποιες αξιολογήσεις αντικτύπου και επίσης πρέπει να υπάρξει και ένα πρόγραμμα εφαρμογής της στρατηγικής πληροφορικής ε, βάση του ΜΑΣΠ που προκύπτει από ε, τα τελωνία 2013 να γίνει μια μελέτη ε, σχέσης κόστους και αποτελεσματικότητας σε σχέση με τον τομέα για παράδειγμα των ειδικών φόρων κατανάλωσης και του ΦΠΑ. Δεν έχει πολύ νόημα αν δεν συμπεριλάβουμε και άλλους έμεσους φόρους κατά τη γνώμη μας. Και ένα τελευταίο σημείο θα πρέπει να γίνει μια μελέτη με, για τη χρηματοδότηση και τους σπόρους που υπάρχουν για τη χρηματοδότηση αυτή. Επίσης θα θέλαμε τέλος να ε, ολοκληρώσουμε λέγοντας ε, ότι η επιτυχής εφαρμογή θα έχει πολύ ε, σημαντική πραγματικά ωφέλη για τα ενδιαφερόμενα μέρη, δηλαδή τα κράτη-μέλη, τους πολίτες, ε, το εμπόριο, αλλά βέβαια επιζητά και τη συμμετοχή των συγκεκριμένων ομάδων, ε, εκτός από τους πολίτες βέβαια. Κάθε ε, άλλη ομάδα πρέπει να συμμετέχει περισσότερο στη φάση της εφαρμογής της όλης διαδικασίας. Και ένα τελευταίο σημείο, ε, μόνο μπορούμε να επιτύχουμε αν υπάρχει σωστή ε, διαχείριση που θα καθοδηγήσει ολόκληρη τη ναι. διαδικασία. Αυτά σε γενικές γραμμές θέλαμε να πούμε. Δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να προσθέσει κάτι από τους συναδέλφους. Ευχαριστούμε. Τάσαμε λοιπόν στο τέλος της παρουσίασής μας και είμαστε διαθέσιμοι για ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Θα σε ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά περιεκτικότατη η περίληψη και που θέτει πολλές ερωτήσεις και ερωτήματα. Δεν είμαι σίγουρος πόσο χρόνο θα έχουμε σήμερα να τα καλύψουμε όλα αυτά. Ίσως υστερότερα, αν ο κύριος Ελίνσκι θέλει να σχολιάσει, θα μπορούσα να του δώσω τη δυνατότητα να το κάνει υστερότερα. Εξ ονόματο τη Γενική Διεύθυνση Επιτροπή. Ε, δεν ήταν δυνατόν να έρθει πιο πριν συνάδελφο. Ε, Μόλι έφτασε. Δεν ξέρω αν κάποιος από του συναδέλφους μου θέλει να αρχίσει με ερωτήσει Για να ξεκινήσω θα ήθελα και εγώ να πω δύο λόγια. Θέλω να σας δώσω κάποια θέματα να αντιδράσετε σε κάποια πολύ σημαντικά ζητήματα. Πρώτα απ' όλα θα έλεγα, πιστεύω ότι οι πολύ μεγάλες διακοιμάνσεις και ε, των καλύτερων ή χειρότερων περιπτώσεων σενάριο μεταξύ 5 ετών και 21 ετών. Το βρίσκω πραγματικά πολύ εκπληκτικό. Υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη διακύμανση, τεράστια διακύμανση. Και όταν κάνουμε λόγο για εξελίξει IT, σε 21 χρόνια για την εξέλιξη τέτοιων συστημάτων, εγώ θα έλεγα 10 γενές, γενές ολόκληρες ε, τεχνολογίας ε, μπορούν να ε, εξελιχθούν. Δεν είναι ρεαλιστικό έτσι να προγραμματίζουμε, θα έλεγα, τουλάχιστον σε μια τέτοια χρονική κλίμακα, διότι διαρκώς ε, θα έχουμε θέματα ε, ενημέρωση επικαιροποίηση. Θα ήθελα να μας ε, εξηγήσετε με δύο λόγια παραπάνω για ποιο λόγο επιλέξατε τέτοιο μεγάλο σενάριο, ευρύ σενάριο για τις καλύτερες και χειρότερες περιπτώσεις. Καλή κίνηση θα ήταν αυτή, διότι θα φώτιζε και άλλα θέματα. Ίσως να ξεκινήσουμε έτσι λοιπόν. Ευχαριστώ. Πραγματικά πρέπει να πω ότι το χρονικό πλαίσιο προκλήθηκε από τις απαντήσεις ε, των εμπλεκόμενων stakeholders. Υπήρξε επιμερισμό σε τρία, σε τρία τμήματα. Νομικές διατάξεις, ε, λειτουργικές διατάξεις, ε, εφαρμογές. Όλα αυτά πρέπει να γίνονται με μια αλληλουχία χρονική. Και σημειώσαμε κατά πόσον οι εμπλεκόμενοι θα θεωρούσαν ότι θα απαιτούσε κάποιο χρονικό διάστημα να γίνει αυτό από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, από τις εθνικές αρχές και για την νομική εφαρμογή, για να ολοκληρωθεί η πρώτη διεργασία, διαδικασία για να ξεκινήσουν όλα αυτά. Ήδη αυτή η φάση θα έπαιρνε από έξι μήνες μέχρι και πέντε χρόνια ως χρονικό πλαίσιο. Αν προσθέσετε επιπλέον άλλα στοιχεία όπως τις τεχνικές εφαρμογές της IT με τεχνικές βέλτιστες προδιαγραφέ που υπάρχουν ήδη για τέτοια συστήματα IT θα μπορούσαμε να πάμε από 5 χρόνια μέχρι και 18 χρόνια διάρκειας συνολικά. Αλλά αυτό τι θα σήμαινε, ότι μετά από αυτή την περίοδο θα είχαμε πλήρη εφαρμογή και υλοποίηση. Φυσικά βέβαια φαίνεται ότι παίρνει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αυτό. Είναι όμως πολύ σύνθετο, περίπλοκο ζήτημα υπό το πρίσμα ότι όλα τα διευρωπαϊκά συστήματα IT μέχρι σήμερα αποκλειστικά σε μια προσέγγιση πελατειακή, πελατών λειτουργούσαν και πρέπει τώρα να διασφαλίσουμε ότι θα μπορούν να αλληλεπικοινωνούν, να ε, αλληλεπικοινωνούν και να μπορούν να καλύπτουν όλες τις προσεγγίσεις όλες δηλαδή τις ε, software, hardware, IT που θα πρέπει να αναπτυχθούν για να καλύψουμε αυτό το φάσμα. Και για να διασφαλίσουμε ότι αυτά θα γίνουν αντιλήπτα, αναφερθήκατε σε σχέση με τεχνολογίες όπως το cloud computing, ολόκληρες συστοιχίες ε, ηλεκτρονικών εγκεφάλων που θα μπορούσαν να διευκολύνουν και να προαγάγουν σε ένα ενιαίο σύστημα. Προς ενημέρωσή σας, ε, έχουμε ζητήσει και μελέτη για κάποιες ε, επιπτώσεις ε, των πολιτικών αυτών των εξελίξεων. Αλλά παρακολουθούμε και εμείς αυτό το τομέα έργα. Για να επανέλθω στο θέμα, δεν είμαι βέβαιος ότι απαντήσατε σε σχέση με τις εξελίξεις των τεχνολογιών, πώς μπορούν τα πράγματα να διαμορφωθούν. Τι μας λέτε, ότι η τεχνολογία μπορεί να εξελιχθεί, να μετεξελιχθεί προς αυτή την κατεύθυνση ή θα έχουμε και ανεδαφικές τεχνολογίες μέσω αυτού του χρονικού πλαισίου. Δηλαδή διασφαλίζει το χρονικό πλαίσιο της τεχνολογίας όσον αφορά τη λειτουργία τους ή καλύπτουμε μια μεταβατική φάση ή μήπως δεν έχουν οριμάσει όλα αυτά. Όλα, λέγει ο μιλητής, θα εξαρτηθούν από την επιλογή της στρατηγικής IT. Όμως ευχαρίστως να να διαβιβάσω αυτό το ερώτημα στον συνάδελφο για τα τεχνολογικά θέματα που είναι παίων επ' παρέμβασή του. Ο λόγος για τον οποίο αναλύσαμε ε, σε σχέση με, προσεγγίσαμε τεχνολογίες όπως το cloud computing είναι σε σχέση με τα, ε, τις στιβάδες ε, τα εφαρμογής και προσέγγισης με, σχέση, σε, με βάση την ταχύτητα. Μετά από τρία χρόνια μπορούμε να έχουμε ακόμα εξελίξεις τεχνολογικές στην τεχνολογική στιβάδα σε σχέση με την ταχύτητα που θα ακολουθείτε σε ένα ή τρία χρόνια με βάση αυτές αυτές τις προσεγγίσεις μπορούμε να έχουμε διαφορετικές, ας το πω έτσι, ταχύτητες από πλευράς τεχνολογιών. Ευχαριστώ. Now, which Άλλες ερωτήσεις, Σμιτ, ε, ε, που φυσικά ήταν, ακούστηκαν επικρίσεις για το γεγονός ε, της καθυστέρησης. Νομίζω δεν ακούσατε την εισαγωγή που αναφέρ, ανέφερε ότι 21 χρόνια θα χρειαστούν, που δεν είναι και πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ, συγγνώμη που άργησα, αλλά είχαμε διακοινοβουλευτικέ συναντήσει στην Επιτροπή Οικονομικών ε, με ε, τα Εθνικά Κοινοβούλια και έπρεπε να παρέμβω και εκεί. Λοιπόν, εγώ διάβασα το χειρότερο σενάριο. Το 2033 εγώ θα έχω πεθάνει το 2033. Τι να σας πω. Μα πώς είναι δυνατό, αυτό είναι το ερώτημά μου. Ίσως θα έπρεπε να θέσω το ερώτημα εδώ, στα αριστερά μου, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τα υπόλοιπα συμφωνώ, αλλά πραγματικά δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για το 2033. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας. Το, το κανονικό σενάριο δηλαδή είναι το χειρότερο σενάριο. Ε, Εμεί λίγο το καλύψαμε αυτό, λέει ο Πρόεδρος, λίγο πριν, πριν έρθετε. Αλλά βλέπω και η κυρία Λιγκρή που θέλει να πάρει τον λόγο. Κύριε Βαλτεσάρη, καλώς ήρθατε. Γιατί είστε και εισηγητής μας στο πρόγραμμα Φίσκους. Αν θέλετε και εσείς να πάρετε το λόγο, ευχαριστώ στο μεταξύ, κυρία Λεγκρίπ Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω ένα ερώτημα. Πέρα από τις δυσκολίες, τεχνικές δυσκολίες που αναφέρθηκαν, που θα δικαιολογούσαν αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα. Ποιο θα ήταν το κόστος για τους ε, καταναλωτές και τους επιχειρηματίες ε, μίας, ενός εξυγχρονισμού των συστημάτων πληροφορικής που χρειάζεται τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι θα μπορούσε... Δεν νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε φάση μεταβατική τόσο μακρά θα έπρεπε να έχουμε στενότερα χρονικά περιθώρια και να αποφασίσουμε ε, ποιες θα είναι οι διορθώσεις, οι δυνατότητες για να γίνει πιο λειτουργικό το σύστημα, πιο νωρίς αυτό το νέο σύστημα. Ευχαριστώ. Το θέμα του χρονοδιαγράμματος και της τεχνολογίας, μήπως μπορείτε λιγάκι να μας το απαντήσετε, μας απασχολεί. Μήπως μπορείτε λίγο περισσότερο να εμβαθύνετε στις ε, απαντήσεις που δώσατε προηγουμένως. Ναι. ξεκινήσαμε με το καλύτερο σενάριο που είναι πέντε χρόνια για αυτή τη διαδικασία εφαρμογής και πήγαμε μέχρι ένα σενάριο πάνω από 20 χρόνια. Αλλά πιστεύουμε ότι μια εφικτή προθεσμία για την εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος μπορεί να μας φτάσει μέχρι το 2020. Γιατί, Γιατί τα υπόλοιπα διευρωπαϊκά συστήματα πληροφορικής δείχνουν ότι έχουμε ήδη τώρα αποκτήσει πολύ πείρα, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε Εξαρτάται βέβαια και από την ε, προσέγγιση πληροφορικής που χρησιμοποιούμε. Αν έχουμε το cloud computing για παράδειγμα ή την τυποποίηση των ε, ε, πλατφορμών σημαίνει ότι θα χρειαστούμε και άλλο χρόνο. Όσον αφορά το κόστος για τους εμπόρους, για τους συναλλασσομένους, δεν έχει ακόμη εκτιμηθεί, δεν το έχουμε υπολογίσει. Γι' αυτό προτείναμε να γίνει μελέτη αξιολόγηση αντικτύπου και σχέσεις κόστους ε, αποτελεσματικότητας, κόστους ωφέλου. πριν αρχίσουμε την εφαρμογή, το πρόγραμμα εφαρμογής ε, της πληροφορικής που προτείνουμε, γιατί τα ερωτήματα που θέσαμε εμεί τους ε, ενδιαφερομένους μας έδειξαν ότι όλα θα εξαρτηθούν από το πόσο θα είναι τυποποιημένα, αν θα είναι κεντρικά ή όχι. Και από 50.000 ευρώ μέχρι 2 εκατομμύρια ευρώ ακούσαμε ποσά. Κανένας λοιπόν δεν έχει κάνει αυτόν τον υπολογισμό. Maybe to add, um, Κατά την άποψή μας, Όλα εξαρτώνται από το αν υπάρχει μια στρατηγική πληροφορικής ε, που να μπορεί να λειτουργήσει. Και αυτά είναι από τα σχόλια που έχουμε για την αναδιατύπωση πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα εργασίας για την πληροφορική. Πρέπει να έχουμε ένα πλήρες ολοκληρωμένο σύστημα πληροφορικής. Αν γίνει κάτι τέτοιο, πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι πολύ μικρότερο το χρονικό διάστημα από το χειρότερο σενάριο. Όχι, δεν είναι το σημείο κίνησής μας το χειρότερο σενάριο. Εμείς πιστεύουμε ότι το 2020 είναι μια λογική ημερομηνία και μέχρι τότε Μέχρι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πει ότι θα τα έχουμε καταφέρει. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό θεωρεί ως ε, εφικτή ημερομηνία. Όχι, μην ξεκινάτε από την ιδέα ότι το 2033 είναι αυτό που εμείς θεωρούμε ως ε, λογική προθεσμία. Και εγώ πέρασα λίγο χρόνο με την ομάδα ε, συζητώντας το συγκεκριμένο αυτό θέμα. Ο λόγος ε, που καταλήξαμε στο 2033 ήταν βάση των εμπειριών που έχουμε από εφιστάμενα συστήματα που πήραν από 6-7 χρόνια 6-7 ε, χρόνια για την ψηφιοποίηση μια συγκεκριμένη διαδικασία. Γι' αυτό ακριβώ ε, σα παραπέμπω στο, ε, στα 10 σημεία τη τελική διαφάνεια παρουσίασή μα που λένε ότι πρέπει να πάρουμε το χρόνο να εξασφαλίσουμε κατά πόσο, να εξασφαλίσουμε ότι ένα κεντρικό σύστημα θα επισπεύσει την κατάσταση. Ε, το cloud computing είναι μια ιδέα. Μπορεί να υπάρχουν και άλλες όμως. Πρέπει να εξασφαλίσουμε, να εξετάσουμε σε βάθος τι θα γίνει, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αν δεν τα κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Ποιο θα είναι το κόστος του να είμαστε πιο αργοί και επίσης ποιο θα είναι το κόστος για την καθημερινή ζωή του πολίτη. Και μιλάμε τώρα για end-to-end management. Γι' αυτό προτείνουμε ε, εκθέσεις ε, από την αρχή της διαδικασίας εφαρμογής μέχρι το τέλος, αλλά να συνεχίσουν οι εκθέσεις και ακόμη μετά το πέρας της εφαρμογής. Μάλιστα. Ο κύριος Φαμπ. Να σας πω την αλήθεια. Εγώ εκπλήσωμαι. Δεν είναι πρώτη φορά που το συζητάμε αυτό το θέμα εδώ. Και εγώ δεν είμαι αυτή τη στιγμή σε θέση να ελέγξω κατά πόσο το cloud computing ή ένα server θα είναι η καλύτερη λύση. Αυτός δεν είναι ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να το αξιολογήσει, να σας πω την αλήθεια. Και πιστεύω ότι είναι λίγο τρελή αυτή η ιδέα. Θα ήθελα να ρωτήσω για τους, ε, τους εμπειρογνώμονες μας ποιος είναι υπεύθυνο ε, για την αποτυχία. Μήπως μπορείτε να μας πείτε είναι αποτυχία το ότι το κράτος μέλος θέλει να, τα κράτη μέλη θέλουν να συνεχίσουν με τα 27 διαφορετικά συστήματα πληροφορικής τους και ε, ε, εθνικούς ε, παρόχους διαφορετικούς. ίσως θα πρέπει να δώσετε μια σαφή καθοδήγηση στα κράτη-μέλη και θα ήθελα πρώτα εσείς να μας δώσετε μια σαφή απάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, συμφωνώ με την ερώτηση του κυρίου Σφάμπ, κύριε Πρόεδρε, αλλά εσείς πιστεύετε ότι είναι συνετό να αναφέρετε ημερομηνία 2033 αν εγώ θέλω να καθυστερώ, να αναβάλω, αν είμαι εθνική αρχή, θα έλεγα, α ωραία, μέχρι το 2033 ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Έχω πάρα πολύ χρόνο. Τι να σας πω, ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορούσε να μας απαντήσει αυτή την ερώτηση, αλλά πραγματικά νομίζω ότι δίνει ένα περιθώριο ελιγμών σε όσους δεν θέλουν να κάνουν απολύτως τίποτε. Βέβαια, η εναλλακτική θα μπορούσε να είναι ότι είναι τόσο σοκαριστικό το 2033 που δεν θα θέλουμε καθόλου να φτάσουμε σε, αυτή τη, σε αυτό το σενάριο. Τέλος πάντων. Να δώσουμε το λόγο και στην κυρία Σκή, η οποία θα θέλει και εκείνη το λόγο. Να απαντήσω. Και θα με συμπληρώσει και ο Ρίτ. Σημαντικό ερώτημα που πήραμε. Θέμα πήραμε, θέλαμε να δούμε το χρονοδιάγραμμα στη μελέτη. Ποια είναι η καλύτερη περίπτωση, ποια χειρότερη. Επειδή λάβαμε υπόψη την χειρότερη περίσταση, δεν σημαίνει ότι αυτό πρέπει να επιλέξουμε, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε γιατί αυτή η χειρότερη υπόθεση θα μπορούσε τελικά να υλοποιηθεί αν δεν προηγηθούν τα αναγκαία οικοδομικά τμήματα που προβλέπει το Κοινοβούλιο για να είμαστε σίγουροι ότι θα εφαρμοστεί το σύστημα ταχαίως. Κάτι που θα ωφελεί τους πάντες και σε καλό κόστος. Να προσθέσω κάτι. The recommendation given within the report. Η συστάση που αναφέρεται στην έκθεση είναι ότι πιστεύουμε το 2020 είναι εφικτή ημερομηνία. Το 2020 ξεκινάει, το 2033. 2020 είναι εφικτός στόχος. Δοθέντως αυτό που είπε είναι ότι θα υπάρχει πλήρες σχέδιο εφαρμογής και μια πάρα πολύ καλή στρατηγική όσον αφορά τα συστήματα πληροφορικής τα οποία χρησιμοποιούνται. Καλοσχεδιασμένη στρατηγική νομίζω είναι σωστή διατύπωση, λέει ο Πρόεδρος. Ο κ. Σβάμπ ρώτησε κάτι. Ποιος είπε ότι είναι υπεύθυνο. αν υπάρχει αντίσταση στα κράτη-μέλη για κεντρικό σύστημα και αν αυτό είναι κρίσιμος παράγον στον οποίο οφείλονται οι καθυστερήσεις. Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα που έθεσε ο κύριος Σβάμπ. Απάντηση. Νομίζω ότι είναι ένα μείγμα. Ο τρόπος λειτουργίας των τελωνιακών αρχών, ο σημερινός, οδηγεί στο να είναι αυτή η υπεύθυνοι οι τελωνιακέ αρχέ και τα κράτη-μέλη όσον αφορά τη λειτουργία του στήματο πληροφορική για την ε, συλλογή των τελωνιακών δασμών. Και κάθε φορά που χρειάζεται αλλαγή ενό συστήματο, χρειάζεται να γίνεται ιδέουσα προσαρμογή 27 κράτη-μέλη. Άρα η διαδικασία είναι πολύ μακρά και συχνά γίνονται παράλληλε διαδικασίε. Παράλληλη διαδικασία δίπλα στην κανονική. Δηλαδή παράλληλα κανονική γραφειοκρατική και παράλληλα ηλεκτρονική. Ποιο ήταν το πρόβλημα. Κανείς δεν μπορούσε να εκτιμήσει, χωρίς ανάλυση, πόσο χρόνο χρειάζεται εφαρμογή κάθε συστήματος πληροφορικής. Δεν έγινε πραγματική έρευνα πάνω σε αυτό. Ούτε έχει ληφθεί κάποια απόφαση για τη στατηγική περιπληροφορικής. και νομικά υπάρχει πρόβλημα. Μάλλον νομικά μπορεί να εφαρμοστεί το σύστημα της πληροφορικής, αλλά τα σύστηματα υποστήριξης θα λείπουν. Όλοι θέλαμε να το εφαρμόσουμε το σύστημα μέχρι το 2013, ήμασταν αισιόδοξοι. Ε, αλλά για να το πω ειλικρινά, χρειάζεται πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να τα καταφέρουμε. Αυτό να φέρουμε και στην έκθεση. Να προσθέσω κάτι. Όπως είπε ο Ντέρκ, έχουμε κράμα, δύο παραγόντων, μείγμα. Κάποια κράτη-μέλη επιμένουν να κρατήσουν το σύστημά τους. Δεν θέλουν να το χάσουν. Ένα στοιχείο αυτό. Άλλο στοιχείο που διαφαίνεται σαφώς από τη μελέτη. Πολλά κράτη-μέλη έχουν προβλήματα λόγω έλλειψης προσανατολισμού από Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουν κάποιο χάρτη, αν θέλετε, πώς να προχωρήσουν πώς να εφαρμόσουν μια στρατηγική για την πληροφορική. Άρα πρέπει να γίνουν επιλογές. Όσο δεν γίνονται επιλογές, δεν προχωράει το πράγμα. Πρόγραμμα εργασίων για την πληροφορική αναφέρει το αναδιατυπωμένο κείμενο. Αυτό είναι κρισίμου σημασία για να, περάσουμε, να ολοκληρώσουμε τη, τη φάση. Καλό σημείο αυτό για να καλέσουμε τον κύριο Ζαλίνσκι να σχολιάσει τα όσα υπόθηκαν μέχρι τώρα και να τον ρωτήσουμε αν θέλει να σχολιάσει κάτι, να θέσει ερωτήσεις προς τους ε, εμπειρογνώμονες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να πω ότι καλωσορίζουμε τη μελέτη. Είναι ποιοτική. Έχουμε προβεί σε μια προκαταρκτική αξιολόγηση. Δεν είχαμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Αρχικά σχόλια έχω σήμερα μόνο. Βασίζονται στην εκτελιστική σύνοψη και στα κεφάλαια 4-5, δηλαδή εξολόγηση και συστάσεις και ελάχιστε ε, προαπαιτήσει, ελάχιστε προδιαγραφέ. Καταρχά. Ήταν ποιοτική προσπάθεια που κατεβλήθηκε την έκθεση. Ζητήθηκε άποψη 8 κρατών μελών. Άρα ατελής η εικόνα που σχηματίζεται. Συνεχίζονται οι συζητήσεις με όλα τα κράτη-μέλη. Και ίσως η τελική εικόνα να είναι διαφορετική. Είδαμε στη διαφάνεια πόσα κράτη-μέλη υποστηρίζουν κεντρική λύση και πόσα μη κεντρική. Δεύτερον, η προθεσμία ημερομηνία ήταν 15 Σεπτεμβρίου 2011. Άλλαξαν πολλά. και συνεχίζονται οι εργασίες με ταχύ ρυθμό. Αναφέρθηκε επανειλημμένα η στρατηγική για την ε, πληροφορική. Έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αυτό, αλλά δεν μπορούμε μόνοι μας να ετοιμάσουμε στρατηγική. Ετοιμάσαμε ειδικέ δομές. Διευθύνουσες ομάδες υψηλού επίπεδου, αναπληρωτών διευθυντών των, των τελωνιακών ε, αρχών. Και αύριο έχουμε τη συνεδρίαση. Το πρόβλημα δεν είναι το όραμα, αλλά η συνεργασία των κρατών μελών για τη στρατηγική. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη και το συμφέρον άλλων εμπλεκομένων, κυρίως του εμπορικού τομέα. Και οι εμπορικοί κύκλοι και αυτοί είναι διχασμένοι. Υπάρχει άλλο θέμα. Τα κράτη-μέλη που διαφέρουν και διαφέρουν και σε μέγεθος μεταξύ τους. Πρέπει Πρέπει να βρούμε μια λύση, μια μέση λύση. Συζητάμε με τα κράτη-μέλη και συζητάμε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρησιμοποιούμε ταυλιτή γεωμετρία στις συζητήσεις μας. Δεν μπορούμε να βρούμε μια γενική λύση. Δημιουργούμε ομάδες κρατών μέλων και εξετάζουμε το ενδεχόμενο, κυρίως ομάδες των μικροτέρων κρατών μέλων. Μπορεί να είναι παρόμοιο το κόστος για μεγάλη και μικρή χώρα, διότι τα σημεία διαπαφής είναι τα ίδια και τα συστήματα είναι παρεμφερή. Και θέλουμε και συστήματα ασφαλείας, δηλαδή να, έχουμε, να, μην, έχουμε περιτά συστήματα. Θέλουμε να έχουμε συστήματα που μπορούν να εφαρμοστούν όχι μόνο από ένα κάτω μέλος, αλλά από πολλά. Άρα να έχουμε εναλλακτικέ λύσεις θέλει να πει ο μιλητή. Τώρα είναι το άλλο θέμα, κεντρική μη κεντρική λύση. Δεν αφορά μόνο την πληροφορική, αφορά την ασφάλεια επίση. Σταθερότητα των συστημάτων. Ευθύνη των διαφορεών φορέων στα διαφορετικά τη κράτη-μέλη. Σας διαβεβαιώ ότι η στρατηγική για την πληροφορική είναι στο επίκεντρο των μελημάτων μας. η 15η Σεπτεμβρίου 2011 δεν ετηρήθηκε. Ετοιμάζουμε τη δεύτερη εκδοχή του σχεδίου του Μάστριχτ. Έχουν πλησιάσει το τελικό στάδιο. Για την τρίτη εκδοχή του βασικού σχεδίου, συγγνώμη, όχι του σχεδίου Μάστριχτ, του βασικού σχεδίου. Και θέλουμε και πολιετές στρατηγικό σχέδιο, το οποίο θα παρουσιαστεί σε μερικές εβδομάδες και στο πολιετέ στρατηγικό σχέδιο θα βάλουμε και το σχεδιασμό της διαδικασίας εκτέλεσης. Όχι μόνο για τον ε, τελωνιακό κώδικα της Ένωσης, αλλά για όλα τα τελωνιακά συστήματα. Δεν βασίζονται όλα τα τελωνία μόνο στον τελωνιακό κώδικα της Ένωσης. Υπάρχουν πάρα πολλές άλλες νομοθεσίες που πρέπει να καλυφθούν από τα συστήματα πληροφορική. Για να μην μακρηγορώ, ολοκληρώνω. Ξεκίνησα λέγοντας ότι καλωσορίζουμε την έκθεση. Όμως, έχουμε κάποιε ερωτήσει. Χρειαζόμαστε κάποιες διευκρινήσει ενδεχομένω. Ανακαλύψαμε και κάποιες εκπλήξεις. Έχουμε επικοινωνία μεταξύ ECS, όχι CTS μόνο, ECS, ICS, έχουμε διάφορα συστήματα άλλα για την επικοινωνία μεταξύ τελειωνικών αρχών. Προς διευκρίνηση. Επαναλαμβάνω τα ήδη υποθέντα. Στην πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε την προθεσμία 2020. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Well, thank you very much. Indeed, indeed... Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε και για την ευκαιρία να υπάρξουν εδώ τοποθετήσεις η κυρία Τεκρυπίνη, η συγγήτρια. Έχετε κάποια άλλα σημεία που θα θέλατε να καλυφθούν. Το Επίτροπο σε μέσα τον καλωσορίζω. Θα γίνει η εισαγωγή αυτή η διεξοδικότητα. Συνέχεια βλέπουμε το ενδιαφέρον σε αυτά τα χατοφυλάκια. Η κυρία Λεγκρίπ, θέλετε να τοποθετηθείτε. Πολύ γρήγορα ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς ζητώ συγγνώμη διότι δεν κατάφερα να έρθω εγκαίρως ε, στην Επίτροπη Ιστορικής Αγοράς και δεν μπορώ να παραστώ στην παρουσίαση αυτής της μελέτης. Ε, Εψήφιζα σε άλλη επιτροπή, αλλά κοίταξα, εξέτασα προσεκτικότατα και εξαντλητικά τους καρπούς των εργασιών αυτών. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τις, προσ... τις προσαρμογές που χρειάζεται να γίνουν στο μέλλον. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έκανε την πρόταση αναδιατύπωσης του εξυγχρονισμού του Ελληνικού Κώδικα την περασμένη εβδομάδα. Είναι καραπός διαφόρων συζητήσεων με του Γενικού Διευθυντέ των Τελωνίων των Κρατών Μελών και διαφόρων, με διάφορου εθνικού εμπειρογνώμονε. Είναι πολύ μακροσκελέ το έγγραφο τεχνική φύσεω, πάνω από 250 σελίδε. Χρειάζεται χρόνο για ενδελεχή ανάγνωση του εγγράφου. Τούτων λεχθέντων. Νομίζω ότι αναφερόμενοι στις ανησυχίες που εξέφρασε το Κοινοβούλιο και στην έκθεση Σαλβίνη για τον συγχρονισμό των τελωνιακών υπηρεσιών, μπορούμε να προωθήσουμε κάποια σημεία. Προφανώς την αναβολή εφαρμογή του ελληνικού κώδικα. Είδαμε από τη μελέτη τα υπαρξιακά θέματα που τίθενται όσον αφορά την ημερομηνία, την νέα ημερομηνία, την αισιόδοξη και την απεσιόδοξη εκδοχή της εφαρμογής του νέου συστήματος πληροφορικής. Άλλο θέμα. Η συνθήκη της Λισαβόνας με τον κώδικα ε, κατά εξουσιοδότηση πράξης και λοιπά, αρμοδιότητες εκτέλεση, υλοποίηση και λοιπά. Αυτά ήθελα να πω. Ε, εκτελεστικές πράξεις, κατεξοδότηση πράξης, εκχώρηση εξουσιών κλπ. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να τα εξετάσουμε. Νομίζω ότι ε, τους επόμενους μήνες ε, και εβδομάδες επανειλημμένα θα μπορέσουμε να επανέρχουμε σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Καλώς. Ευχαριστώ την ομάδα Cooper που ήρθε εδώ και μας παρουσίασε σαφέστατα το θέμα. Πραγματικά σημαντικός πόρος για την κυρία Λεγκρίπ και τους κύριους τον κύριο Σμπαντεσάρη, εξετάσει το πρόγραμμα Φίσκους, διότι είναι περίπλοκο, δύσκολο θέμα και αυτή η Επιτροπή μάλιστα είναι νέα σε αυτό το θέμα. Ξεκίνησε η όλη εξέλιξη πριν το 2009. Αυτή είναι, αυτό είναι το πρώτο σημαντικό στοιχείο που πρέπει να εξετάσουμε εμείς. Έγιναν διάφορες παρουσιάσεις ήδη. Και ευχαριστώ τον Ζελέσκη, την ομάδα του και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με το θέμα αυτό. Πολύ χρήσιμο έγγραφο αυτό μαζί με την πρώτη Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Επιτροπής που όπω ακούσατε υιοθετήθηκε 10 Φεβρουαρίου θαρώ. Οπότε σύντομα θα έχουμε το κύμα μπροστά μα, Η κυρία Λεγκρίπ είναι ε, η συγγήτριά μας που ασχοληθεί με το θέμα και νομίζω ότι θα είναι πολύ άσχολη τι επόμενη μήνε η κυρία Λεγκρίπ αλλά προσβλέπουμε στην πρόθεση του όλου θέματο. Λοιπόν, αυτά για εκείνου που μα βλέπουν από το διαδίκτυο και πολλοί στα τελωνία ενδιαφέρονται. Αυτό το έγγραφο θα διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μα, οπότε θα μπορέσετε να το κατεβάσετε και να διαβάσετε την έκθεση με την ησυχία σα. Και σίγουρα, και στρέφομαι στην κυρία Λεγκρίπ, θέλουμε να επανεξετάσουμε κάποια στοιχεία των λογογράφου και ίσω να καλέσουμε κάποιου από την ομάδα PricewaterhouseCooper για να συζητήσουμε δελεχέστερα μαζί με την ομάδα τη ηγήτρια το ζήτημα. Και θα θέλαμε να ακούσουμε και ποιε θα ήταν οι παρατηρήσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν θα είχα την καλοσύνη να μα στείλετε τι παρατηρήσει, θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμε. Καλώ. Οπότε μπορούμε τώρα εγκαίρω να καλωσορίσουμε τον Επίτροπο κύριο Σεμέτα στην σημερινή μα συνεδρίαση και το πλαίσιο τη συναντήσεω είναι το εξή. Ξεκινάμε, συνάδελφοι, μια σειρά συναντήσεων με επιτρόπους οι οποίοι καλύπτουν το τομέα εργασιών της Επιτροπής στα πλαίσια του διαθρωμένου διαλόγου για το 2012 να μας πούνε ποιο είναι το πρόγραμμα εργασιών τους. Και νομίζω ότι τα θέματα τα οποία θέλουν να προωθήσουν στο προσωρινό τους πρόγραμμα εργασιών το 2013 και 2014. Διότι όπως νομίζω ξέρει η Επίτροπος, η Επιτροπή μας αρέσκεται στο να εξετάζει με στατηγικό τρόπο αυτά που κάνουμε και γι' αυτό να θέσαμε και μια μελέτη πριν λάβουμε τις προτάσεις σας διότι από πέρσι τον Ιούνιο ξεκίνησαν εργασίε σε αυτό το τομέα, οπότε ήδη ουσιαστικά προηγούμεθα του προγράμματος εργασιών σας, ακολουθούμε τον των προτέρων το ρυθμό σας. Θα θέλαμε όμως να με συνημερώσετε σχετικά με αυτό και άλλα θέματα τα οποία θα θέλετε να μας ε, θέσετε και μετά θα ακούσετε ερωτήσεις από τα μέλη. Λοιπόν, καλώς ήρθατε για μία ακόμη φορά και με τα να σας δώσω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Πολλά συνέβησαν από τελευταία μου επίσκεψη και ανταλλαγή απόψεων μαζί σας σε αυτή την Επιτροπή. Τα τελωνιακά θέματα σας είναι πασίγνωστα και εντυπωσιάζομαι από την μεγάλη ποιότητα, υψηλή ποιότητα των συζητήσεων και των εκθέσεων. Όπως ε, ήδη το συζητήσαμε στην έκθεση Σελβίν, ε, κάνατε και άλλη μια συζήτηση για την εφαρμογή του εξεχωρισμένου τελωνιακού κώδικα επί τη βάση μιας μελέτης που θα δώσει χρήσιμες πληροφορίες και περαιτέρω προβληματισμούς. Σκοπός μου σήμερα είναι διτός. Πρώτα απ' όλα να ανταλλάξω απόψη μαζί σα για πρόσφατε πρωτοβουλίε που προτάθηκαν και να σα ενημερώσω δεύτερον για πρόσφατε εξελίξει και για το πρόγραμμα εργασιών για το 2012. Επειδή ο χρόνο είναι περιορισμένο, θα σα δώσω μια σύντομη επισκόπηση. Μάλλον μια σύντομη επισκόπηση σα έχει μοιραστεί εκ των προτέρων όσον αφορά τι πρωτοβουλίε που έχουν δρομολογηθεί. Αφήστε με λοιπόν να ξεκινήσω αναφερόμενος στα θέματα που βρίσκονται στα χέρια των συνομοθετών. Όπως αναφέρθηκε το, την περσινή άνοιξη, έχουμε βάλει μια πρόταση για την αδιάθρωση του εξυγχρονισμού του ελληνικού κώδικα που θα καλείται ο τελωνιακό κώδικα Ένωση από τούδε και στο εξή. Δεν επισέτω σε λεπτομέρειε τη προτάσεω αυτή καθεαυτή, αλλά δράτω με τη ευκαιρία για να ενθαρρύνω του συνομοθέτε να περιορίσουν το εγχείρημα τη αναδιατύπωση στα αυστηρό αναγκαία. Και να μην μπείτε στον πειρασμό να ανοίξετε το κουτί της Πανδώρας και τους ασκούστε όλου ε, και τον όσο συμφωνήθηκαν στην περίοδο διαπραγματεύσεων 2005-2008 είναι κοινό συμφέρον να τελειώσει αυτός ο πρώτος γύρος το εξυγχρονισμό του ελληνιακού κώδικα, τη διαδικασία εξυγχρονισμού, τόσο ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την επόμενη φάση. Εν την προετοιμασία των επομένων κεφαλαίων, διενεργούμε μία αξιολόγηση της Τελωνιακής Ενώσεως για να μπορέσουμε να βρούμε ποια κενά υπάρχουν, ποιες ανάγκες υπάρχουν σε αυτό το πλαίσιο. Πολλοί από τους προβληματισμούς σας που εκφράστηκαν στην έκφραση Σολβίνη χρήζουν περαιτέρω προσοχή. Πρώτα απ' όλα θα ακολουθήσουν σωστή σειρά. Πρώτα απ' όλα, θέλετε να διευκολυνθεί η υιοθέτηση της ανδιατύπωσης του ελληνικού κώδικα πριν από την προθεσμία της 24ης Ιουνίου του 2013. Αυτό είναι κάτι που ε, απαιτείται. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, το σχέδιο εφαρμογής είναι φιλόδοξο αλλά αξιόπιστο και απαιτεί πλήρη δέσμευση και προσπάθεια όλων των μπλεκομένων φορέων και όσον αφορά την τεχνογνωσία και όσον αφορά την ε, χρηματοδότηση της τεχνολογίας πληροφορικής. Αυτό αναφέρεται και στη μελέτη που σας παρουσιάστηκε μόλις τώρα. Η προτινόμενη προθεσμία της 21ης Δεκεμβρίου του 2020 βασίζεται επί της υποθέσεως ότι τέτοια δέσμευση μπορεί να εξασφαλιστεί. Το πρόγραμμα Φίσκους έχει σχεδιαστεί να προσφέρει την αναγκαία υποστήριξη. Χαίρομαι, συνεπώς, που με πληροφορούν ότι το έργο για το Φίσκους θα ξεκινήσει σύντομα με τον κύριο Μπαλτεσάρη. Πρόσφατα διορίστηκε συγητή. Αυτό θα πρέπει να μα βοηθήσει να θετήσουμε το νέο πρόγραμμα ιδεοδό μέσα του 2013. Το ΦΙΣΚΟΥΣ έχει σαν στόχο την υποστήριξη τη Ελληνική Ένωση και την ενίσχυση τη εσωτερική αγορά, βελτιώνοντα τη συνεργασία μεταξύ των τελωνιακών και φορολογικών αρχών, κυρίω μέσω τη αναπτύξεω και συντηρήσεω διευρωπαϊκών συστημάτων πληροφορική. Το νέο πρόγραμμα βασίζεται στα ισχυρά σημεία φυσταμένων προγραμμάτων εισάγοντα μόνο περιορισμένε αλλαγέ. Η βασική αλλαγή είναι η συγχώνευση του τελωνιακού και του φορολογικού προγράμματο, των τελωνιακών και φορολογικών προγραμμάτων. Ποια είναι η λογική που ακολουθήσουμε, να απλουστεύσουμε και να εξοθολογήσουμε τα δύο προγράμματα στο ευρύ πλαίσιο των πολιετών δημοσιονομικών πλαισίων. Γνωρίζω ότι γίνονται προσπάθειες από κάποιες αντιπροσωπείς στο Συμβούλιο να διαχωριστεί το φίσκους σε δύο ξεχωριστά προγράμματα. Κατά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τέτοια κίνηση θα έστενε τα λάθο μηνύματα προ του πολίτε, δηλαδή ότι οι συνομοθέτε έχουν κολλήσει σε μια προσέγγιση λανθασμένη και αρνούνται απλουστεύσει και εξορθολογισμό. Λοιπόν, βασίζομαι σε εσά να υποστηρίξετε την συγχωνευμένη αυτή πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελα να στραφώ σε πολύ επίκαιρο θέμα για την ΙΜΚΟ, την εφαρμογή των δικαιωμάτων των πνευματικών από πλευρά τελωνίων. Με τα χαρά βλέπω πόσο εντατικά έχετε εργαστεί όσον αφορά την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αύριο θα ψηφίσετε την έκθεση του κυρίου Κρόιτσμαν, οπότε θα ήθελα να πω κάποια λόγια σχετικά με τον μελλοντικό κανονισμό. Καταρχά, βασίζομαι στην υποστήριξη του Κοινοβουλίου για να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογή των παραβιάσεων πνευματικών δικαιωμάτων που καλύπτονται από τον κανονισμό. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει εκ των προτέρων κάποιο λόγο να συμπεριλάβουμε κάποια πνευματικά δικαιώματα και να αποκλείσουμε κάποια άλλα Όπω είναι το παράλληλο εμπόριο από πλευρά τελωνιακή προστασία, όλα τα πνευματικά δικαιώματα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και θα πρέπει οι τελωνιακέ αρχέ να αποφασίζουν πώς θα εστιάζουν τις δραστηριότητε τους λαμβάνοντας υπόψη ε, τους σχετικούς κινδύνους. Συνεπώς πιστεύω ότι ο κανονισμός θα επιτρέπει στις τελωνιακέ αρχές να δρουν επί σαφών περιπτώσεων παράνομου παράλληλου εμπορίου. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέχει τις αντιδράσεις που δημιουργεί η απόφαση του δικαστηριού για την Nokia Philips για την ε, διαμετακόμιση παρανόμων αγαθών μέσω της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει προσφέρει την καλύτερη λύση για την αντιμετώπιση του θέματος μετακόμιση και τώρα και στο μέλλον. Εδώ δεν υπάρχει τον προτέρων λόγος για να περιορίσουμε το πεδίο εφαρμογής των, ε, της παρεμβάσεως των ελληνικών αρχών στη διαμετακόμιση. Η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν σαφής. Ο κανονισμός για τις αρχές είναι διαδικαστικός κανονισμός και όχι ένας κανονισμός που καθορίζει τα ουσιαστικά ε, τα δικαιώματα. Θα πρέπει ε, η ουσιαστική νομοθεσία να καλύπτει και η νομολογία του δικαστήριου το θέμα της διαμετακόμισης. Δεν μπορούμε να καθορίσουμε πνευματικά δικαιώματα από την πίσω πόρτα μέσω του τελωνιακής νομοθεσίας. Είναι θεμελιώδες θέμα θα πρέπει εμείς σε μια παγκόσμια αγορά να αφήσουμε να περνάνε ελευθέρως κάποια αγαθά μέσω της επικρατής Ευρωπαϊκής Ενώσεως χωρίς την άδεια του δικαιούχου. Στο ουσιαστικό δίκαιο για πνευματική νομοθε... ε, ιδιοκτησία θα το εξετάσουμε. Ο τελωνικό κανονισμό δεν θα πρέπει να εξυπηρετεί αυτό το σκοπό. Θα πρέπει να επιτρέπει όμω μελλοντικέ εξελίξει όσον αφορά αυτό το βασικό δίκαιο, ουσιαστικό δίκαιο. Τέλο, ελπίζω ότι ο μελλοντικό κανονισμό θα διατηρεί ε, τις δυνατότητες που έχουν τα τελωνία να μέσα στον τομέα και να είναι φτηνό το κόστο. Ε, θα πρέπει να πληρώνει ο κάτοχος των δικαιωμάτων το κόστο τη τελωνιακή εφαρμογή. Αν δεν εξασφαλίζεται αυτό δεν θα κινούνται πλέον τα τελωνία. Η ευθύνη άλλων φορέων όπω είναι οι μεσάζοντες είναι εκτό του πεδίου εφαρμογή του κανονισμού για τα τελωνία. Προσβλέπω σε μια επιτυχή ολοκλήρωση των συζητήσεων επί του κανονισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και ελπίζουμε να ολοκληρωθεί επί δανεικής προεδρίας της Ευρωπαϊκή Ένωση σύντομα να μπορεί να ωφεληθεί από ισχυρότερη εφαρμογή των μέτρων προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων πλευρά τελωνίων. Να στραφώ τώρα για τις εξελίξεις όσον αφορά τον τομέα της ασφάλειας και των διεθνών σχέσεων. Σε σχέση με τα εκρηκτικά και σφαίρες από την Ιεμένη, σε σχέση με την εμπλοκή της διεθνούς κοινότητας και άλλους εμπλεκόμενους στη διεθνή αλυσίδα ανεφοδιασμού, δείχνει ότι πρέπει να τελούμε εγρηγόρση όσον αφορά τους κινδύνους που εγκυμονούν. Είχαμε τελωνιακέ οργανώσεις που πέρσι τόνισαν την διάχυση και πρόοδο όσον αφορά τέτοιου είδους στοιχεία πριν από τη φόρτωση αεροσκαφών προχωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την προετοιμασία νομοθετικού έργου που θα μπορέσει να ολοκληρώσει τον τελωνιακό κώδικα ώστε να υπάρχει η βελτίωση της διαθεσιμότητας και των, της ποιότητας στοιχείων τέτοιας ε, έγκαιρης προειδοποίησης. Αυτό θα δίνει τη δυνατότητα να συμπληρώνουν οι τελωνιακές αρχές ε, τις προσπάθειες ε, των αρχών ασφάλειας αεροπορικών μεταφορών. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη επίσης και το βιομηχανικό περιβάλλον και έχουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Εξπρεσέ να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτές τις αρχές ε, όσον αφορά και την νομοθετική διαδικασία από κοινού με τους, ε, τις ταχυδρομικές αρχές ε, και την ομάδα πραγματογνωμονών που δημιουργήθηκε για να καλυφθούν οι ανησυχίες για την ασφάλεια όσον αφορά την αποστολή αντικειμένων ιδιαίτερα όσον αφορά την Οικουμενική Σύνοδο στην Τόχα αυτών των εμπλεκομένων το Σεπτέμβριο 2012. Στον παγκοσμιοποιημένο σημερινό κόσμο για το εμπόριο πρέπει να βασιζόμαστε σε πολυμερείς δράσεις καθώς και σε διμερή τελωνιακή συνεργασία. Αυτό με φέρνει στις διεθνείς ε, δεσμεύσεις μας, ε, ιδιαίτερα όσον αφορά και τους ε, ανατολικούς γείτονες και τους κυριότερους εμπορικούς εταίρους της ΕΠΑ και την Κίνα σημαντικές εμπορικές ροές ε, διασταυρώνουν τα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να ενταθεί η συνεργασία με τους ανατολικούς εταίρους ώστε να υπάρξει η σωστή διαχείριση των κινδύνων. Κινδύνων όσον αφορά την ε, παράνομη διακίνηση αγαθών. Δύο συμπληρωματικές προσεγγίσει προτείνω. Πρώτον, διμερώς να συμφωνήσουμε σε στρατηγικά πλαίσια που θα ταυτοποιούν προτεραιότητες αμοιβαίου συμφέροντος με συγκεκριμένες δράσεις και προγράμματα εφαρμογής και λειτουργίας. Αυτό έγινε με την Κίνα, Ρωσία και την Μολδόβα. Η Ουκρανία είναι η επόμενη χώρα σε αυτή την προσέγγιση. Η δεύτερη προσέγγιση στο επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, το λαθρεμπόριο των προϊόντων καπνού, διότι αυτό είναι επιβλαβές για την κοινή αγορά. Και έτσι έχουμε υποβάλει ένα συνολικό πρόγραμμα δράσης που θα εμπλέκει και τους ανατολικούς εταίρους στη δράση. Τώρα πρέπει να έχουμε πλήρη δέσμευση από όλους όσους εμπλέκονται για να αντιμετωπιστεί αυτού του είδους η απάτη. Τώρα η μετάθεση προς τα δυσμά ε, της ε, προσοχής μας για την ένταση της διατλαντικής συνεργασίας όσον αφορά τα θέματα ασφάλειας. Και πέρσι τον Ιούνιο, Επίτροπος Μάνστον και εγώ υπογράψαμε ένα τέτοιο πλαίσιο υπέρ της ασφάλειας αποκινούμε Τζανέτ Ναπολετάνο τον ΙΠΑ. Αυτό τοποθετεί και θέτει την τροχιά των κοινών συμφερόντων και κοινή δράσης πολυμερός και διμερός η διατλαντική αυτή προσπάθεια εξελίσσεται σε διαφορετικούς άξονες. Πρόοδος ε, συνήθει όσον αφορά την αμοιβαία αναγνώριση ε, των προγραμμάτων εταιρικής σχέσης ΕΕ και ΕΠΑ. Μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση διαπραγματεύσεων μας πέρσι τον Νοέμβριο, η αμοιβαία αυτή αναγνώριση την Άνοιξη θα προσυπογραφεί και έτσι θα υπάρχει η πιστοποίηση για την ασφάλεια που θα ξεκινήσει να λειτουργεί από τον Ιούλιο και εφ' Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας ενεργά εμπλεκόμεθα στην νομοθεσία που ακολουθούν οι για την 100% σάρωση εμπορευματοκιβωτίων. Η Υπουργός Αναπολετάνο είπε ότι τον Μάιο το αργότερο θα δώσει τη δυνατότητα επέκτασης κατά δύο έτη τη προθεσμία του Ιουλίου. Έχουμε και συμπληρωματικέ προσπάθειε ε, των αρχών τη ε, ΕΠΑ ώστε να προωθηθεί νομοθετικό έργο στο Κογκρέσο. Η στρατηγική που πρόσφατα υιοθετήθηκε όσον αφορά την ασφάλεια επιβεβαιώνει ότι η σχέση αυτή από πλευρά ΕΕ και ΕΠΑ για ένα πολυμερέ πλαίσιο ακολουθεί αυτή την πολυμερή δράση και όχι την μονομερή προσέγγιση και δράση. Συζητώντα με την ε, Υπουργό Ναπολετάνο τον, Ναπολετάλο τον Νοέμβριο 2011, συμφωνήσαμε να εντείνουμε τη συνεργασία μα όσον αφορά την ασφάλεια των αερομεταφερόμενων φορτίων. Θα έχουμε και μια αντιπροσωπεία μα που θα μεταβεί στη ΣΥΠΑ ώστε να συζητηθεί το πώ η ΕΠΑ ΕΕ και η ΕΕ μπορούν να συνεργαστούν στο πλαίσιο της ε, προηγμένη προηγμένης αυτής σάρωσης εμπορευματοκιβωτίων από πλευράς ΣΥΠΑ. ΕΕ. Όσον αφορά την Κίνα, τις εμπορευματικέ ροές θέλουμε να τις ε, ε, θέσουμε σε ένα πλαίσιο με ε, διευρυμένη διεθνή συνεργασία με την εφαρμογή των ρητρών IPR, της ασφάλειας και των περιορισμών που πρέπει να ακολουθούνται όσον αφορά την αντιμετώπιση των απατών. Η IPR είναι προτεραιότητα. Τα στατιστικά στοιχεία όσον αφορά τα, τις τελωνιακές αρχές δείχνουν ότι 85% των αγαθών προέρχονται από την Κίνα το νέο πρόγραμμα δράσης ε, ΚΙΝΑ ΕΕ που ξεκίνησε το 2009 έδωσε κάποια αποτελέσματα ήδη και είναι φυσικά ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα με ένα μακροπρόθεσμο χρονορίζοντα και έτσι θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας με την Κίνα για να σημειωθούν σημαντικές πρόοδοι στο μέλλον στον τομέα της ασφάλειας όσον αφορά την ε, προσφορά και ζήτηση συνεχίζουμε τις ε, δράσεις μας με πιλωτικά προγράμματα και σε σχέση με την ασφάλεια τελωνιακών αρχών και προδιαγραφών. Επίσης εξετάζουμε την ε, φυκτότητα το δυνατόν να υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση τέτοιου είδους προγραμμάτων μεταξύ ΕΕ και Κίνας. Το κύριο συμφέρον μας είναι να προαχθεί η διάχυση αυτών των στοιχείων όσον αφορά τους εταίρους μας στην Κίνα και να ενισχυθεί η διαχείριση κινδύνων μέσω αμοιβαία τέτοια προσέγγιση από πλευρά των Κινέζων, Κινέζικων αρχών. Και όσον αφορά τις ΗΠΑ, Κίνα και την ανατολική μας πολιτική για τους ανατολικούς γείτονες, θέλουμε να προαγάγουμε την ημερήσια διάταξή μας σε οποιασδήποτε επαφές και ε, διαβουλεύσεις θα γίνονται. Τώρα, σε σχέση με τα κυριότερα χαρτοφυλάκια τα οποία ε, προανέφερα, προσβλέπουμε στο να ακούσουμε τις απόψεις σας ε, που θα είναι προς όφελός μας από πλευρά της Κοινοβουλευτικής σας Επιτροπής στο Ευρωκοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πίτροπε για μια πολύ χρήσιμη και πάρα πολύ περιεκτική ε, παρουσίαση. Μας ενημερώσατε και για κάποιες διεθνείς δραστηριότητές σας παρά το γεγονό ότι μας ενδιαφέρουν όλο ιδιαίτερω αυτές που αφορούν την παραχάραξη. Οπότε, ερωτήσεις τώρα. Όποιος ε, μου απέσπασε την προσοχή πρώτος, δεν ξέρω αν κανείς άλλος θέλει να πάρει το λόγο. Mr. Mr. Mr. Schwab and Mrs. Uh, and Mr. and Mr. Αυτό ήταν ο κατάλογος των ομιλητών. Έχουμε χρόνο. Δεν θέλω βέβαια να, χάσω το λόγο να, να μην δώσουμε τη δυνατότητα για απάντηση στο τέλος, οπότε να ακούσουμε κάποιους, ε, κάποιες ομάδες ερωτήσεων και μετά να υπάρξει απάντηση. Οι δύο πρώτοι ομιλητές. Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Γκάλ Πέλτς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα εισαγωγικά σας σχόλια. Είναι πολύ σημαντικά τα ζητήματα αυτά βέβαια και είναι και πολύ σημαντικά για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την ε, κοινή ενιαία και εσωτερική αγορά. Έχω μια γενική ερώτηση θεωρητικής φύσεως και θα ήθελα να με βοηθήσετε να διαφωτιστώ. Έχω ασχοληθεί με την, τον προγραμματισμό της φορολόγησης ε, και με έχει απασχολήσει το θέμα θεωρητικά και πρακτικά. Αν εμείς λοιπόν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια εσωτερική ενιαία αγορά, αυτός είναι ο στόχος όλων των κρατών μελών και φαίνεται ότι η ίδρυση, η δημιουργία της αγοράς αυτής είναι ε, προς όφελος των κάποιων κρατών μελών ε, επειδή θα είναι ιδιαίτερα υποφελής για αυτά, όμως κάποια κράτη-μέλη ε, θα είναι σε μειονεκτική θέση λόγω της αγοράς αυτής. Ένα από τα μέσα της αγοράς είναι η φορολογική πολιτική, η οποία βέβαια για την ώρα είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών είναι ένα ε, εργαλείο της οικονομικής πολιτικής. Οι φορολογικές αλλαγές λειτουργούν και έτσι ε, υπέρ μιας ομάδας ε, συμφερόντων και κατά μιας άλλης ομάδας συμφερόντων. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι πάρα πολύ απλό. Γνωρίζετε φορολογικές αλλαγές ή φορολογική πολιτική που δεν προβαίνει σε διάκριση ή εν πάση περιπτώσει δεν επιφέρει αλλαγές στον ανταγωνισμό έχετε λάβει υπόψη σας ότι η πτυχή από τη, η οπτική γωνία από την οποία βλέπουμε τα πράγματα μήπως θα έπρεπε να είναι διαφορετική γιατί βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι εξετάζει τα πράγματα αλλά αν ο στόχος μας ο κύριος είναι να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης και να δούμε κατά πόσο θα επιτύχουν αυτό το στόχο τα κράτη-μέλη δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη ότι πηγαίνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι μια βασική, μια θεμελιώδης προσέγγιση. Αν δεν ολοκληρώσουμε το ζήτημα αυτό, αν δεν το επιλύσουμε δεν μπορούμε να μιλάμε για την νέα αγορά ούτε για τη φορολογική πολιτική. Ευχαριστώ. Ναι, πραγματικά είναι μια ευρύτατη ερώτηση, όχι μόνο για τον κύριο Σεμέτα, αλλά και για άλλους. Η κυρία Σολτιμούζα. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε, που προσήλθατε και συμμετείχατε σε αυτόν τον πολύ σημαντικό διάλογο μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρώτα, μια ερώτηση θα είχα Μιλήσατε για την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων όσον αφορά θέματα ε, τελωνιακά κτλ. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας για το θέμα της άκτα. Πώς η άκτα θα αναμειγνύεται και θα παρεμπλέκεται σε σχέση με αυτό το πεδίο, σε αυτό το θέμα. Το Κοινοβούλιο θα απασχοληθεί με την άκτα τους επόμενους μήνες. Θα ήθελα την άποψή σας για αυτό το πεδίο για αυτό το θέμα. Μετά είπατε ότι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να πληρώνουν όσον αφορά τα έξοδα ε, τελωνιακά και άλλα για την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων. Συμφωνούμε με αυτό. Θα ήθελα να ακούσω όμω την άποψή σα για την ασφάλεια σε σχέση με τα προϊόντα. Αν συμφωνείτε πράγματι με το ότι θα πρέπει να είναι οι αρχέ εκείνες που είναι υπεύθυνε για να διασφαλίζουν ότι προϊόντα εισερχόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι ασφαλή. Από κοινού με και του παραγωγού. Παρ' όλα αυτά, πάλι ελπίζω θα συμφωνείτε ότι είναι ευθύνη των κρατών μελών να διασφαλίζουν ότι θα είναι επίσης ασφαλή αυτά τα προϊόντα. Έχετε κάποια επισκόπηση συνολικά, μια άποψη τι γίνεται από πλευρά των κρατών μελών, πώς χρηματοδοτείται αυτή η ασφάλεια των προϊόντων, αυξάνεται, βρίσκεται σε ευθύνουσα πορεία, τι συμβαίνει. Ελπίζω ότι θα υπάρχει σωστή αντίδραση γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ε, Uh, Ευχαριστώ πολύ. Σε σχέση με το πρώτο ερώτημα, ελπίζω να το κατάλαβα καλά. Πρέπει να πω ότι εμείς πιστεύουμε ότι ο συντονισμός της φορολογικής πολιτικής Ευρωπαϊκή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαδραματίζει πολύ σημαντικότερο ρόλο και οι ενέργειες Ευρωπαϊκής Επιτροπής κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Δείτε για παράδειγμα την τελευταία μας έρευνα για την ετήσια ανάπτυξη. Έχουμε λάβει υπόψη μας τη συνιστόσα τη φορολογική ως τμήμα της έρευνας αυτής και αυτό δείχνει ότι ο συντονισμός της φορολογικής, των φορολογικών πολιτικών ε, αποτελεί πλέον ε, αναπόσπαστο τμήμα του ευρωπαϊκού μας εξαμήνου. Και άμα δείτε για παράδειγμα ε, τις ε, πρωτοβουλίες μας τις περσινές, προσανατολίζονται όλες προς την καλύτερη, ε, τον καλύτερο συντονισμό της φορολογικής πολιτικής και όλες ασχολούνται με το θέμα των αδυναμιών του φορολογικού συστήματος όσον αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή της, ε, ε, της ε, φορολογικής πολιτικής. Για παράδειγμα, η φορολόγηση της ενέργειας, ε, ε, η οι πρωτοβουλίες μας για τον χρηματοπιστωτικό τομέα όλα, ότι αυτό πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να προσαρμόσουμε την ε, ε, προσέγγιση μας αυτήν και να λάβει το ε, Συμβούλιο τις απαραίτητες αποφάσεις το συντομότερο δυνατόν. Θέσατε και το θέμα της φορολογικής απάτης. Είναι μια βασική προτεραιότητα του προγράμματός μου φέτος και τις ερχόμενες ημέρες ε, θα αρχίσουμε και δημόσια διαβούλευση για την ε, ε, αποφυγή της διπλής φορολόγησης. Ιδέες δηλαδή πώς να καταπολεμήσουμε φορολογικούς παραδείσους και περιορισμούς φορολογικούς που δεν μας διευκολύνουν. Υπάρχουν λοιπόν πρωτοβουλίες σε επίπεδο ένωσης και υπάρχουν και συντονιστικές ενέργειες στις οποίες ήδη έχουμε προβεί και τις εφαρμόζουμε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Όλα αυτά εγώ τα θεωρώ εξελίξεις που είναι πλήρως συμβατές με την καλύτερη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και συμφωνώ Απολύτω ότι η φορολογική πολιτική είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της αποτελεσματικότητας της ενιαία αγοράς και είναι κάτι που πρέπει να εξεταστεί πολύ προσεκτικά. Όσον αφορά το ερώτημα, τα, τα ερωτήματα για την άκτα. Η άκτα από μόνη της δεν αλλάζει το ουσιαστικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, αφορά μια ε, σημαντικότερη συνεργασία των κρατών μελών ε, που συμμετέχουν στην καταπολέμηση των, της, των παραβιάσεων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Επίσης, έχει κάποια στοιχεία ε, τελωνιακής προστασίας, όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη και το πολιτικό κλίμα. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από το δικαστήριο να γνωμοδοτήσει από αυτού. Δεν θέλω εγώ τώρα βέβαια να προκαταβάλω την άποψη του δικαστηρίου, αλλά ελπίζω ότι θα είναι θετική. Σε σχέση με την άκτα. όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων. Συμφωνώ ότι είναι ένα σχετικό καινούριο, αλλά πολύ σημαντικό στοιχείο ε, στην ε, τελωνιακή δραστηριότητα και το τονίζουμε πολύ περισσότερο. Πέρσι, μάλιστα, εγκρίναμε ένα, ένα πακέτο κατευθυντηρίων γραμμών ε, πολύ περιεκτικό σε σχέση με την ασφάλεια των προϊόντων ε, στις ε, τελωνιακές αρχές, κάτι το οποίο επικρότησαν, επικρότησε ιδιαίτερα ο κλάδος και υποστήριξε μάλιστα και επί τη βάση αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών εμείς πιστεύω ότι έχουμε πολύ πιο ομοιογενή προσέγγιση ε, από πλευράς τελωνίων σε σχέση με την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ασφαλείας προϊόντων. Τα τελωνία είναι το πρώτο σημείο ε, στο οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των ανασφαλών προϊόντων ώστε να μην μπουν καθόλου στην αγορά. Γιατί αν αρχίσουν να διανέμονται στις αγορές, το πρόβλημα γίνεται πολύ χειρότερο. Γι' αυτό ακριβώς δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ε, δραστηριότητα αυτή των τελωνιακών μας αρχών. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι η κυρία Καλπέτς θέλει να πάρει και πάλι το λόγο, να δευτερολογήσει από αυτού, αλλά δυστυχώς ε, πρέπει και άλλοι να λάβουν το λόγο. Αν έχουμε χρόνο στο τέλος θα σας ξαναδώσω το λόγο. Κανιέτε και Κομφεράτη. Ε, ε, Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ για τις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις. Θα ήθελα να αναφέρω στο ερώτημα για τις, την καλή λειτουργία των ε, τελωνίων. Από την Λετωνία προέρχομαι, μια συνοριακή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεματοφύλακα επίσης προστάτη των εξωτερικών συνόρων της ε, Ένωσης. Η ασφάλεια των συνόρων, αν δούμε τώρα τις συνθήκες, είναι σαφές και αναφέρεται σαφώς. Νομίζω είναι η 325 παράγραφος ότι κάθε κράτος μέλος πρέπει να διασφαλίζει τα δικά του οικονομικά συμφέροντα εξίσου όπως διασφαλίζει και θα διασφαλίζει τα ενωσιακά οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ένα από τα κύρια μέσα γι' αυτό είναι η αποτελεσματική καλή λειτουργούσα διαδικασία των τελωνίων, σύγχρονα τελωνία και διαδικασίες και υπηρεσίες για, μια, για συνοριακές χώρες να εξυγχρονίσουν τις ε, τελωνιακές τους υπηρεσίες απαιτεί πολλές ε, μεγάλα κονδύλια σε χρηματοοικονομικές επενδύσεις. Και αν δούμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον προϋπολογισμό 2014-2020, υπάρχει ένα πρόγραμμα φίσκους προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό το πρόγραμμα δεν διαθέτει και δεν διασφαλίζει επιπρόσθετη χρηματοοικονομική αρρωγή στις συνοριακές χώρες. Δεν θα ήταν όμως προς όφελος και προς το συμφέρον όλων των κρατών μελών να γινόταν αυτό οι μεθοριακές, οι συνοριακές χώρες να μπορούν να έχουν πρόσθετη αρρωγή χρηματοοικονομική συνδρομή για την, τον εξοπλισμό και καλύτερη λειτουργία των τελωνίων τους από τον ίδιο τον προϋπολογισμό, τον ενωσιακό. Θα είσαστε πρόθυμος να γίνει κάτι τέτοιο, να εγκριθεί μια τέτοια πρόταση στο μέλλον υπέρ αυτών των χωρών. Και στρέφομαι στον πρόεδρο για να ολοκληρώσω τώρα, στον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής, επειδή δεν αισθάνομαι ευχάριστα να μην μπορώ να μιλήσω τη γλώσσα μου. Επειδή η λετωνική γλώσσα είναι η επίσημη, μια επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν είναι η πρώτη φορά που δεν μπορώ να έχω αυτή την υπηρεσία και να χρησιμοποιήσω τη γλώσσα μου. Και είμαι υποχρεωμένη να χρησιμοποιώ μια γλώσσα εκτός της μητρικής μου γλώσσας. Ευχαριστώ. Thank you. I'll, I'll respond to, to your point. Λοιπόν, θα απαντήσω αργότερα σε αυτό που είπατε. Ο κύριος Κονφεράτη έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, εσείς μας είπατε ότι είσαστε υπέρ μιας λύσεως που θέτει μαζί την Τελωνιακή Ένωση με τη Φορολογική Ένωση. Μας εξηγήσατε για ποιους λόγους κάνετε μια κοινή πρόταση Κυρίως πολιτικά στοιχεία αναφέρατε ότι πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα στους Ευρωπαίους πολίτες και γι' αυτό θέλετε, θέλετε να είναι όσο πιο ενωμένο γίνεται το μήνυμα και να δώσει κάποια ανάσματα. Εσείς και οι συνεργάτες σας δεν αξιολογήσατε αντικειμενικά ποιε είναι οι δυσκολίες ενός μόνο νομοθετήματος γιατί είναι δύο τομείς, δύο θέματα που αναμφισβήτητα έχουν κάποια στοιχεία διασύνδεσης αλλά και έχουν μεταξύ τους διαφορετικές δυναμικές συνθήκες που επικρατούν. Και αν αυτά τα στοιχεία της διαφοράς, άσχετα με τις διασυνδέσεις τους που, έχουν, που θα έχουν στο τέλος διαδικασίας, αν αυτά τα στοιχεία της διαφοράς, μήπως θα έπρεπε να εξεταστούν, να αντιμετωπιστούν μέσω δύο διαφορετικών νομοθετημάτων. Οι δύο τομείς να παραμείνουν χωριστοί. Γιατί το ρωτάω αυτό διότι ανησυχώ. Φοβάμαι ότι η όλη δυναμική των δύο τομέων είναι διαφορετική. Και η διάσταση, το βάρος που απορρέει από τη διασύνδεση ίσως μας κάνουν να χάσουμε όχι μόνο χρόνο, αλλά να χάσουμε και την εμβάθυνση και την ανάλυση που θα μας επέτρεπε ξεχωριστή προσέγγιση με διαφορετικά νομοθετήματα. Φοβάμαι ότι τελικά θα έχουμε μια πολύ γενική προσέγγιση, διότι θέλουμε να κρατήσουμε μαζί πράγματα που εξ αρχή είναι απόμακρα μεταξύ τους. Αυτό το ερώτημα ήθελα να θέσω. Το σκεφτήκατε αυτό. Κάνατε αυτή την ανάλυση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό ήθελα να θέσω ένα ερώτημα και σα ευχαριστώ. Επίτροπε. Well, regarding... Σε σχέση με τις ε, μεθοριακές μας ε, χώρες, ε, τις χώρες με τις οποίες συνορεύουμε ειδικότερα προς Ανατολάς. Καταλαβαίνω ότι λέτε και γι' αυτό πέρσι πρότεινα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για τις χώρες αυτές ε, της Ανατολικής Ευρώπης και μέσω κοινών δράσεων αλλά και μέσω τεχνικών, ε, τεχνικής υποστήριξης αλλά και πολλών άλλων δραστηριοτήτων για να, μπορέσουν ε, να, να μπορέσει να ενισχυθεί η προσπάθειά τους, η δυνατότητά τους να, να υποστηρίζουν, να προστατεύουν τα σύνορά μας. Από οικονομικής απόψεω. Υπάρχει το πρόγραμμα Φίσκους που ήδη είναι ένα βήμα προς τα εμπρός γιατί προβλέπει κοινή εργασία όσον αφορά την ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής, οπότε είναι πολύ σημαντικό και θα δώσει τη δυνατότητα οικονομιών μεγάλων στα κράτη-μέλη, γιατί θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε ένα κοινό σύστημα πληροφορική, το οποίο μετά θα μπορέσουμε να το μοιραζόμαστε μεταξύ κρατών μελών. Αυτό είναι ο στόχο του προγράμματο FACECUS. Όσον αφορά τώρα τον εξοπλισμό, οι χώρες με τις οποίες ανα, ε, συνορεύουμε ανατολικά μας έχουν ε, ζητήσει εξοπλισμό, σαρωτές ή άλλου είδους ε, εξοπλισμό στο πλαίσιο των ε, ταμείων περιφερειακής ανάπτυξης επίσης ε, μπορούμε να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν. Έχουμε συζητήσει, ίσω και διαπραγματεύσει θα μπορούσαμε να τι αποκαλέσουμε με τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειών, πώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια αυτά για τελωνιακούς σκοπούς. Και πώς μπορούμε να το προβλέψουμε στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι τα κράτη αυτά πρέπει ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια αυτά για να μπορέσουν να συμμετέχουν στην προστασία των ε, συνόρων των ανατολικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά σε σχέση με τα προβλήματα που αναφέρατε. Όσον αφορά το πρόγραμμα φίσκους τώρα, κατά πόσο θα πρέπει να είναι ένα ή δύο προγράμματα, αν κατάλαβα καλά το ερώτημά σας. Συζητήσαμε πολλές φορές ε, τα ωφέλη δύο προγραμμάτων ε, και τις αρνητικές ε, επιπτώσεις που θα μπορούσαν να υπάρχουν και καταλήξαμε στην κοινή παρουσίαση γιατί υπάρχει ανάγκη ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ φορολογικών και τελωνιακών αρχών και δυστυχώς δεν ισχύει πάντοτε αυτό σήμερα. Συγχωνεύουμε δηλαδή τα προγράμματα σε ένα, αλλά από την άλλη υπάρχουν ε, συγκεκριμένες ε, διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των φορολογικών και των τελωνιακών ζητημάτων. Και προτείνουμε μία λύση νομίζω που από τη μία απλοποιεί το σύστημα προγραμματισμού και από την άλλη επιτρέπει συνέργειες μεταξύ φορολογικών και τελωνιακών αρχών. Επιπλέον εξασφαλίζει το ότι ζητήματα τα οποία είναι ε, ξεχωριστά για τα τελωνία και ξεχωριστά για τα, τη φορολογία μπορούν ε, να εξεταστούν στο, πρόγραμμα του, του στο, πλαίσιο του προγράμματος διαφορετικά. Ξέρω ότι είναι ζητήματα που σας απασχολούν και εσάς στην Επιτροπή, στην Επιτροπή σας, αλλά πρέπει να λάβετε υπόψη ε, την ε, γενική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία υποστηρίξατε κιόλας, ότι πρέπει να μειώσουμε το περίπλοκο του πολιετούς δημοσιονομικού προγραμματισμού, να μειώσουμε τον αριθμό των προγραμμάτων, να απλουστεύσουμε τα προγράμματα και εμείς προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία που έχουμε για την απλοποίηση του συστήματος. Ενδεχομένως ο κύριος Σάρι να μας ε, πει ορισμένα πράγματα για το θέμα αυτό, μια και είναι εισηγητής. Θα γίνει κοινή εξου, ε, κοινή ε, εξέταση του, προγρα... του θέματος αυτού με την Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή. Καταλαβαίνω τι είπε η κυρία Καλνιέτη για τη διερμηνία. Κάνουμε ό,τι μπορούμε κάθε φορά να λάβουμε υπόψη τα αιτήματα, αλλά βλέπετε ότι είναι ένας μικρός αριθμός διερμηνε... ε, ε καμπίνων διερμηνίας. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ δύσκολο για μένα να εκφραστώ όπως πρέπει σε μια ξένη γλώσσα στη συγκεκριμένη ορολογία. Και αν δεν μπορούσα να μιλήσω καθόλου αγγλικά, πώς θα συμμετείχα στις εργασίες της ε, Επιτροπής μας. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Um, now, then I have Mr. Schwab. και η κυρία Κοράτσα είναι η επόμενη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε που ήρθατε να μας μιλήσετε και να συζητήσετε μαζί μας. Ε, θα ήθελα να αναφέρω τέσσερα σημεία σε αυτά που αναφέρθηκαν για την άκτα. Πρώτα απ' όλα. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι ο κύριος Κρόιτσμαν πραγματικά ε, στην έκθεσή του ε, ασχολείται πολύ με την άκτα. Δεν μπορούμε να πούμε σαν Ευρωπαίοι ότι με τα πνευματικά δικαιώματα ε, τα πνευματικά δικαιώματα είναι θεμελιώδη δικαιώματα και έχουν θεσπιστεί έτσι. Η αξιολόγηση και η προστασία των ε, πνευματικών δικαιωμάτων είναι εθνικό θέμα. Εθνικές αρχές, οι τελωνιακές, ε, που θα εφαρμόζουν την άκτα, αυτοί θα πρέπει να προστατεύουν τα δικαιώματα. Ανεξάρτητα από το που ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα, αν ανήκουν ιδιωτικέ εταιρείε είτε όχι. Και η διεπαφή μεταξύ όλων αυτών είναι ότι αυτά που λέει για τα δικαιώματα είναι ότι θα πρέπει να συμφωνούν οι εταιρείε των πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά η κατάχρηση, η πειρατεία, η παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων είναι κάτι που αφορά και τις θελωνιακές αρχές και αυτό είναι σημαντικό, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίε και κύριοι, όπως είπε και ο πρώην Πρόεδρο Hans Gert Pettering είναι ένα μέρο στον κόσμο όπου δεν είναι αυτός σκοπό η εξουσία και η δύναμη. Και όσον αφορά το 100% της άρρωσης των εμπορευματοκιβωτίων που εισάγονται από ΗΠΑ και αλλού. Το συζητήσαμε στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς ότι δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί ο κώδικας των τελωνίων πριν το 2020. Ε, είναι δύσκολο αυτό. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα δικά μας προβλήματα Ποια είναι τα προβλήματα. Κάποια κράτη-μέλη που είναι μικρά έχουν διαφορετικά συμφέροντα. Όσον αφορά την επεξεργασία εισαγωγών-εξαγωγών. Διαφέρει η αντιμετώπιση τους από ότι στα μεγαλύτερα κράτη-μέρη. Οι μεγαλύτερες χώρες θέλουν μια αγορά ε, και να ακολουθούν τις επιταγές Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής Ένωσης. Τέλο πάντων, ίσω πρέπει να τεθούν κάποια παραδείγματα όσον αφορά την ε, βελτιωμένη συνεργασία. Τρίτον, κάτι που σχετίζεται με παρελθούσε εργασίε. Είπα ότι η ελληνική πολιτική συνδέεται στενά με τη φορολογική. Ισχύει αυτό. Χρειάζεται πιο καλό συντονισμό των πολιτικών αυτών για την ενιαία αγορά. Κυρίω και για τη διακυβέρνηση εσωτερική αγορά. Για να είμαστε ειλικρινεί, σε κάποιε περιπτώσει αμφιβάλλω το κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πρόθυμη ή έτοιμη να μπει στη μάχη που σας χρειαστεί για να περάσει τις πολιτικές που κατευθύνονται προς την ενιαία αγορά. Στην ετήσια έκθεση στην ανάπτυξη δεν ξέρω τι συμπεριλαμβάνεται από τούδε και στεξής. Η κυρία Κοράτσα Μπίλτα έχει κάτι να πει πάνω σε αυτό. Μετά, ο κύριος Κάμπος μόλις απεχώρησε και ο συγγητή για το ηλεκτρονικό εμπόριο, την ομάδα εργασία για το ηλεκτρονικό εμπόριο απουσιάζει. Εκεί είχε υποθεί σε αυτή την ομάδα ότι χρειάζεται ενοποίηση όσον αφορά του κανόνε ΦΠΑ. Χρειάζεται απλούστευση του διασυνοριακού εμπορίου. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά θέλω να ακούσω κάποια πράγματα πάνω σε αυτό. Η ε, κυρία Κοράτσα Μπίλτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, Πέρσι το Κοινοβούλιο ψήφισε μια έκθεση για αποτελεσματικότερη και δικαιότερη ε, πολιτική στον αφορά το λιανεμπόριο στην Ευρώπη. Σας είχαμε ζητήσει να εξετάσετε το θέμα των ε, ειδικών φόρων στην Ουγγαρία. Και εκφράσαμε ανησυχίες, διότι από ό,τι καταλαβαίνουμε η φορολογική πολιτική είναι εθνικό θέμα. Αλλά θέλουμε να έχουμε μια καλά λειτουργούσα εσωτερική αγορά και να σεβαστούμε ε, το δικαίωμα ελεύθερης εγκατάστασης κάθε εταιρείας. Ξέρουμε ότι θέλετε να απαντάτε τα ερωτήματά μας, υπήρξε ανταλλαγή επιστολών, είσαστε σε επαφή με τις Ουγγρικές Αρχές. Ασχοληθήκαμε και εμείς στην Επιτροπή αυτή, συζητήσαμε τον αρμόδιο Υπουργό και στην αντιπροσωπεία της ΣΥΜΚΟ στην Ουγγαρία πέρσι μας είπε η Ουγγρική Κυβέρνηση ότι είναι χρονικά περιορισμένος φόρος και θα με αυτό το 2012. Μιλάμε για ειδικό φόρο επί λιανεμπορίου. Εγώ ανήκω σε εκείνους που πιστεύουν ότι ιδιαίτερα τώρα θα πρέπει να δούμε ότι είναι επιδεινούμενη η οικονομική κατάσταση στην Ουγγαρία, αρνητικό το κλίμα και δεν ενδείκνυται να επιτίθεται κανείς κατά, ενό, κατά ενός κράτους μέλους. Είναι πιο επικοδομητικό για την επίτευξη αποτελεσμάτων να έχουμε εύρυθμα σε εσωτερική αγορά και να συνεχιστεί ο διάλογος. Καλό και για μας και για την ευρωπαϊκή επιχειρηματική κοινότητα. Στο διάλογό μας με τους επιχειρηματίες το τονίσαμε ότι πρέπει να διατηρηθεί ο διάλογος Δεν θέλουμε να υπάρχουν πιο ακρεφνείς και μεγαλύτερος εθνικισμό στην Ευρώπη. Ερώτηση. Τι γίνεται όσον αφορά το διάλογο σας με την Ουγγαρία. Τι κάνετε. Βλέπετε κάποια δυνατότητα να ακολουθούνται ε, διακριτικές πρακτικές που σας οδηγήσουν σε διαδικασίες κατά παράβαση για παραβίαση κάποιων κανόνων. Συνήθως ε, δέχομαι περισσότερες ερωτήσεις για φορολόγηση. στο τελευταίο ερώτημα να απαντήσω. Ολοκληρώνεται η αξιολόγηση του φόρου στην Ουγγαρία. Οι υπηρεσίες μας εξετέλεσαν τεράστιο έργο. Ανέλησαν κάθε λεπτομέρεια του φόρου αυτού στο λιανεμπόριο. Δεν μπορώ σήμερα να σας πω ποιο θα είναι το τελικό πόρισμα. Οι υπηρεσίες θα οδηγηθούν στη θέση την τελική και το πόρισμα. Τελική απόφαση την άνοιξη θα ληφθεί, πιστεύω. για την απλούστευση των κανόνων ΦΠΑ. Πέρσι, όπως ξέρετε, εκδώσαμε ανακοίνωση για το μέλλον του ΦΠΑ. Εκεί καθορίσαμε τις μελλοντικές μας εργασίες στον τομέα. Πρέπει να σας πω ότι η Δανική Προεδρία έχει δραστηριοποιηθεί ιδιαίτερα στον τομέα αυτό. Πρόθεσή της είναι να ετοιμάσει συμπεράσματα του Συμβουλίου με βάση την ανακοίνωση αυτή. Βάσει των συμπερασμάτων θα επικεντρώσουμε τις προσπαθίες μας. Αλλά και χωρίς να περιμένουμε τα συμπεράσματα, προβλέπονται ήδη κάποιες αποφάσεις για φέτος. Παραδείγματος χάρη. Θα ετοιμάσουμε την τον ιστότοπό μας, την πύλη μας στο διαδίκτυο, όπου εκεί θα εμφανίζονται όλα τα ποσοστά ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις. Έτσι, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να εφαρμόσουν σωστά το ΦΠΑ. Φέτος επίσης θα ετοιμάσουμε τριμερή ομάδα θα συμμετέχουν οι επιχειρήσεις, οι φορολογικές αρχές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκεί θα συζητούνται βασικά θέματα που είναι σημαντικά για τις επιχειρήσεις. Διότι ΦΠΑ είναι περιπλοκότατο ζήτημα, πολύ τεχνικό. Είναι σημαντικότατο να ακούμε και να λαμβάνουμε υπόψη τις απόψεις των επιχειρήσεων. Αυτή η τριμερής λοιπόν ομάδα θα είναι το βήμα εντός του οποίου θα γίνεται ανταλλαγή απόψεων. Φέτος επίσης θα ασχοληθούμε με την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ. Θα προτείνουμε μηχανισμό ταχείας αντιδράσεως για νέου είδους απάτες. Αυτές οι δράσεις ήδη προβλέπονται για φέτος. Τα επόμενα χρόνια, 2013-2014, θα υποβάλουμε προτάσεις και άλλες ιδέες που συμπεριλαμβάνονται στις ανακοινώσεις μας για το μέλλον του ΦΠΑ. Και βέβαια η μείωση του διοικητικού άχθους και η απλούστευση είναι βασικό κομμάτι των προσπαθειών μας. Όσον αφορά το συντονισμό των φορολογικών και το AGS. Παρουσιάστηκαν ιδέες. Αυτές του AGS αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες. Όσον αφορά τον συντονισμό της φορολογικής πολιτικής, θα έχουμε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο τέλος της εβδομάδας και ελπίζω ότι αυτές οι ιδέες θα εγκριθούν από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Αυτό θα μας δώσει πλήρη εντολή για να εφαρμόσουμε αυτές τις ιδέες μέσω συγκεκριμένων συστάσεων απευθυνομένων προς τα κράτη-μέλη. Ήδη επεξεργαζόμαστε συστάσεις για φορολογική πολιτική για να απευθύνουμε προς τα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό μέσο για καλύτερο συντονισμό της φορολογικής πολιτικής. Κυρίως όταν μιλάμε για μετακίνηση του φόρου από, τα, από, την, από τις παραγωγικές διαδικασίες προς πιο φιλικές μορφές. Κάποια είδη φορολόγησης ε, όπως τις ε, είναι πιο μετάβλητα και πιο εύκολα μετακινηθούν από ότι άλλες μορφές. Τώρα, όσον αφορά τη δουλειά που κάνουμε, τα δικά μας καθήκοντα και την ανάγκη να κάνουμε αυτό που πρέπει. όσον αφορά την εφαρμογή του εξυγχρονισμένου τελωνιακού κώδικα. Πρέπει να πω σαφώς ότι όπως είδα στην έκθεση της Price Water Coopers ότι υπάρχουν κάποιες αισιόδοξες απεσιόδοξες προθεσμίες. Σας ανιστοιχούν οι απεσιόδοξες προβλέψεις. Η απεσιόδοξη ημερομηνία. που ίσως φύγει και ημερομηνίε που ίσως να μην υπάρχουμε ακόμα πλέον εμείς. Ίσως εσείς να υπάρχετε, ναι. Έγινε προσεκτική αξιολόγηση όταν προετοιμάζαμε την αναδιατύπωση και η προτινόμενη ημερομηνία της αναδιατύπωσης 1η 12 του 2020 είναι ρεαλιστική πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι δεν αφορά μόνο την Ευρωπαϊκή Επίτροπη το θέμα. Αν εξαρτάται από εμά, πιθανότατα θα θα τάχιστα. Εμπλέκονται όμως όλα τα κράτη-μέλη και το σημαντικότερο και τους εμπορικούς κύκλους. Άρα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς δύνανται να εφαρμόσουν τα προβλεπόμενα στον εξυγχρονισμένο τελωνιακό κώδικα. Και, και στην έκθεση Pricewater House Cooper που έκανε προτάσεις και προς αυτή την Επιτροπή που θα διαβαστούν και στο Συμβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα σας ενημερώνει τακτικά για τις εξελίξεις. Έτσι θα γίνει σωστός χειρισμός, ο βέλτιστος δυνατός χειρισμός της όλης διαδικασίας. Ευχαριστώ. Πέντε λεπτά μας έχουν μείνει Σμιτ και Μπαλτασάρη. Και, μετά ο Επίτροπος. Mm, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, Νομίζω ότι είστε πάρα πολύ δραστήριο σε σχέση με την ε, φορολογία και μάλιστα μερικέ από τι προτάσει σα παρά είναι δραστήριε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν πειράζει. Αυτό το συζητήσουμε σε μια άλλη επιτροπή. Ποιο είναι το δικό σα χειρότερο σενάριο για τον εξυγχρονισμένο τελωνιακό κώδικα. Εδώ μας είπαν 2033. Ε, Εσεί τι ημερομηνία μα δίνετε. Ναι, αυτό είναι το ερώτημά μου. Ναι. Εκτός μικροφώνου, Πρόεδρος. Δυστυχώς δεν ακούμε. Η απάντηση πάντως είναι ναι. Έχω και άλλο ερώτημα σε σχέση με την άκτα. Για ποιο λόγο τώρα το στέλνει στο δικαστήριο για να γνωμοδοτήσει το θέμα αυτό. Γιατί δεν το κάνατε πιο πριν εφόσον τη είχαμε ήδη υπογράψει. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπαλτασάρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Φυσικά ευχαριστώ τον Επίτροπο για αυτή τη δυνατότητα συζήτησης κυρίως γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να συνέλθουμε από την απεσιοδοξία που έπιασε την Επιτροπή μας αφού ακούσαμε την ημερομηνίες εφαρμογής του ενημερωμένου, του εξυγχρονισμένου του ελληνικού κώδικα. Οι ερωτήσεις μου είναι δύο. Τα δικά μας σύνορα δεν είναι αδιαπέραστα. Ε, κυρίως όσον αφορά τις πλαστογραφίες γεωργικών ε, προϊόντων και εμπορικών προϊόντων. Αντίθετα μάλιστα οι, οι μεγάλοι χειριστές των, ε, των αυτών, των πλαστοποιημένων προϊόντων των γεωργικών έχουν θύρες εισόδου, χώρες εισόδου πολύ καλά επιλεγμένες ξέρουν ακριβώς σε ποιες χώρες υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή επί κάποιων προϊόντων και σε ποιες χώρες αντίθετα αυτή η προσοχή είναι μικρότερη. Λοιπόν, πώς θα καταφέρουμε σε μια έτσι ολιστική Τελωνιακή Ένωση, όπου το επίπεδο της προσοχής θα πρέπει να είναι ίσο παντού, να εγγυηθούμε ότι υπάρχει το ίδιο επίπεδο προσοχής. Δεύτερη πτυχή αφορά το πόσο σκόπιμη είναι αυτή η πρόταση Ευρωπαϊκή επιτροπή που θεσπίζει το πρόγραμμα δράσης στο κοινό, διότι φυσικά τα επιχειρήματα που μας παρουσιάσατε είναι επιστικά. Όμως οι συνομιλητές μας να είναι οι τελωνιακές ε, αρχές και οι φορολογικές αρχές που θα συνομιλούν για το πρόγραμμα φίσκους. Όσον αφορά τα τελωνιακά θέματα, υπάρχει μεγαλύτερη ενοχή, διαθεσιμότητα, ισοσελαστικότητα από πλευράς κατών μελών, ε, που δεν το βλέπει κανείς τόσο πολύ στα φορολογικά θέματα, που ισχύει εκεί ο νόμος της ε, ομοφωνίας. Η στόχη του προγράμματος είναι διτός, διαφορετική στόχη δύο υποδιαιρεί το πρόγραμμα σε δύο τμήματα. Υπάρχει η ίδια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που ήδη στην πρόταση εμπεριέχει το σπόρο μιας διποδιέρεσης. Το φίσκους μπορεί να διαμορφωθεί με δύο τρόπους. Είναι το, πρόγραμμα, εργασιών διαφορετικό για τον ελληνικό τομέα και για τον φορολογικό τομέα και προβλέπονται ε, δύο συστήματα πληροφορικής διαφορετικά. Εγώ φοβούμαι ως εισηγητής ότι οι δύο καταστάσεις, η φορολογική πτυχή λόγω περιπλοκότητας, λόγω μεγαλύτερης ευαισθησίας που έχει το θέμα αυτό, για τα κάτι μελη μπορεί στο τέλος να καθυστερήσει τη διαδρομή, τη συνολική όλου του προγράμματος και αυτό θα ήταν πραγματικά κρίμα, επιζήμιο. Uh, Πρώτα απ' όσον αφορά την γραμμή αυτή από πλευράς μας. Αυτό που είναι σημαντικό πιστεύω είναι η αναδιατύπωση της πρότασης να εγκριθεί το δυνατόν ταχύτερα η νέα πρόταση αυτή. Πρώτη αυτή η προθεσμία από την οποία θα ξεκινήσουμε τον υπολογισμό των άλλων ε, προθεσμιών και πιστεύω ότι για την ημερομηνία που προτάθηκε σχετικά στην αναδιατύπωσή μας 1η Δεκεμβρίου δηλαδή 2020 που είναι αυτή αλλά επίσης προτείνουμε τα συστήματα να αρχίσουν κλιμακούμενα να εφαρμόζονται και να λειτουργούν δεν σημαίνει αυτό ότι όλα θα πρέπει να αναβληθούν μέχρι το 2020 θα έχουμε κλιμακούμενη εφαρμογή ανάλογα με χώρες. Είναι μια ρεαλιστική ημερομηνία πιστεύουμε και συνεργαζόμενοι από κοινού μπορούμε να συμμορφωθούμε και να την τηρήσουμε. Αυτή είναι η προσέγγιση μας σε σχέση με τους εταίρους μας που και εκείνοι σε αυτό το πρόγραμμα θα μπορούν να ανταποκριθούν στα αιτήματα, στις απαιτήσει αυτές όσον αφορά την ημερομηνία, καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής του κώδικα. Και μετά όσον αφορά το θέμα της άκτα, απόφαση του σώματος, συλλογικού σώματος ε, των επιτρόπων ήταν και έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να προσαρμοστεί και να συμμορφωθεί ανάλογα με την ομολογία και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και σε σχέση με τις ε, συστάσεις ε, του δικαστηρίου όσον αφορά τις υποανάληψη δράσης και τα λοιπά και σε σχέση με το, με το πρωτογενές δίκαιο δεν θα πρέπει να πούμε ότι αλλάζει το νομοθετικό πλαίσιο αυτός λόγω της άκτα. Δεν αναμενόταν να δημιουργηθεί μια τέτοια αντίδραση σε σχέση με την πρόταση αυτή. Όσον αφορά στη συνέχεια το θέμα μιας περισσότερο ενιαίας εφαρμογής όσον αφορά τον δασμολογικό κώδικα, τελωνιακό δασμολογικό κώδικα, αν δείτε τις δικές μας προτάσεις και αν δείτε επίσης προτάσεις που θα υποβάλουμε σύμφωνα φυσικά με το πρόγραμμα που προβλέπετε, όλες στοχεύουν και προσανατολίζονται σε μια πιο ομοιογενή εφαρμογή των κανόνων και κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα τελωνία, τις υπηρεσίες τελωνίων και ο κανονισμός για την εφαρμογή IPR όσον αφορά τις τελωνιακές υπηρεσίες στοχεύει μια πιο ενιαία, ενιοποιημένη εφαρμογή όσον αφορά όλες τις διατάξεις του. Και γι' αυτό πιστεύω ότι από αυτό αυτόν τον κανονισμό, αυτός ο κανονισμός από κοινού με προτάσεις επίσης που πρόκειται να υποβληθούν κατά τη διάρκεια του έτους 2012 όπως την ανακοίνωση για τη διαχείριση κινδύνων και την ασφάλεια όσον αφορά την, ε, ε, τη ζήτηση και την, θα καταστήσει τη διαχείριση αυτών των κινδύνων πολύ, σε ένα πολύ πιο ενιαίο πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα οδηγήσει σε μια πιο ενιοποιημένη εφαρμογή τελωνιακά από πλευράς Ένωσης. Και στόχος μου είναι να καταφέρουμε οι τελωνιακές υπηρεσίες να καταφέρουν να τα βγάλουν πέρα με αυτόν τον τρόπο σε σχέση με τις εφαρμογές κανόνων και κανονισμών που πιο ενιαία θα πρέπει να επιτυγχάνεται η εφαρμογή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, σε σχέση με τα δύο προγράμματα αυτά έναντι ενός, ήδη έχω υποβάλει τα επιχειρήματά μου σχετικά. Φυσικά η συζήτηση μόλις ξεκινά σε σχέση με την κοινοβουλευτική σας επιτροπή για αυτά. Είμαστε πρόθυμοι να προσερχόμεθα και να συζητούμε σε κάθε λεπτομέρεια όλες τις πτυχές αυτού του προγράμματος. Πρέπει επίσης να δούμε και τις εξελίξεις σίγουρα. Ποιες θα είναι οι εξελίξεις στα κράτη-μέλη. Και σε κάποια κράτη-μέλη βλέπουμε ουσιαστικά την συγχώνευση ε, φορολογικών υπηρεσιών και τελωνιακών υπηρεσιών για αυτό. Τέσσερι χώρες δεν θα ήταν καθόλου πρόβλημα να υπάρχει ένα ενιαίο πρόγραμμα και μπορεί σε άλλα κράτη-μέλη αυτές οι εξελίξεις να ακολουθήσουν υστερότερα ως τεκτενόμενα, ως γεγονότα. Είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να συζητήσουμε, κύριε Ισήγητα, αυτό το θέμα μαζί σας για αυτό το πρόγραμμα και να σας υποβάλουμε και να σας παρουσιάσουμε όλα τα επιχειρήματα τα οποία έχουμε. Ευχαριστώ. Ήταν πολύ ενδιαφέρον ότι η έκθεση Pricewaterhouse ε, αναφέρθηκε στα πλαίσια του εξυγχρονισμού του ελληνικού κώδικα στο ότι και εμπλεκόμενοι θα ήθελαν εναρμόνιση τη συλλογή του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωση. Και αυτό ήταν επίση κάτι που αναφέρατε στι σκέψει σα. Κύριε, κύριε Κέπχαρτ, τελείωσε ο χρόνο μα. Θέλει να επανέλθει η κυρία Γκέπχαρτ. Αν μείνετε λίγα λεπτά μετά, μπορούμε διμερό ίσω να συναντηθείτε διμερό και να ακούσετε τι έχει να σα πει διότι τώρα έχουμε περάσει το χρόνο μας κατά πέντε λεπτά και θέλω να ευχαριστήσω τους διερμηνείς για τη δουλειά τους που έκανα το πρωί και να σε ευχαριστήσω και εσάς που ήρθατε ε, και παρακολουθείτε τη συνεδρίασή μας. Είναι πολύ χρήσιμη, ανταλλαγή επίκαιρη, ε, ανταλλαγή απόψεων. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που κάνετε, όχι μόνο για τους τομείς που κάνετε στον τομέα αρμοδιοτήτων, αλλά στο ευρύτερο έργο που κάνετε για του φόρους, πως βλέπουμε στη συνεχιζόμενη συνεργασία μαζί μα και χαίρομαι που αναφερθήκατε στι συστάσει τη εκθέσεω Pricewaterhouse για τακτικέ ενημερώσει του Κοινοβουλίου όσον αφορά τον εξυγχρονισμένο τελωνιακό κώδικα και είναι κάτι που θα καλωσορίζαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και προσβλέπουμε σε συνεχή συνεργασία μα του επόμενου μήνε. Σα ευχαριστώ. Λοιπόν, διακόπτουμε κυρίε και κύριοι μέχρι τι 3 όταν ο Επίτροπος Αλμούνια θα έρθει. Ελπίζω να είσαστε ακριβώ εδώ στι θέσει σα, διότι θα είναι μια ιδιαίτερη περίσταση αυτή να ακούσουμε τι θα γίνει για την πολιτική ανταγωνισμού. Ευχαριστούμε και καλή σα όρεξη.